να ξεκινήσουμε το επόμενο σημείο, με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Να καλωσορίσω τον Υπουργό Πέτερ Πλάσαν, Υπουργό Παιδείας, Επιστήμης, Έρευνας και Αθλητισμού της Σλοβακίας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα αυτά για μας, κύριε Υπουργέ. και στα σχετικά θέματα που θα συζητηθούν επί Ολλανδικ... ε, Προεδρίας είναι το πρόγραμμα πλαίσιο 7 και ο ορίζοντας 2020. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια ενδιάμεση αναθεώρηση γιατί το, το, για το FP7 πρόκειται για μια ε, έκθεση εφαρμογής ενώ και για τον ορίζοντα 2020 μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι πρόκειται για μια ενδιάμεση ε, αναθεώρηση. Επίσης, περιμένουμε την στρατηγική για το διάστημα της Κομισιόν και προετοιμάζουμε το ένατο πλαίσιο πρόγραμμα γιατί σε 1,5 χρόνο θα ξεκινήσουμε την εκπόνηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027. Από αυτή την άποψη λοιπόν χαιρόμαστε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ που είστε μαζί μας. Κύριε Πλάφτσαν. Και θα θέλαμε να κάνετε μια εισήγηση για να ξεκινήσει η συζήτηση. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Yes. Yes. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, πρόσκληση να παρευρεθώ εδώ. Είναι μεγάλη μου τιμή να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του διαστήματος, της επιστήμης και της έρευνας. Χαίρομαι επίσης που σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τις φιλοδοξίες της Σλοβακικής Προεδρίας όσον αφορά την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών θεμάτων και αξιών και την ενίσχυση της συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους τομείς. Παρότι η Σλοβακική Προεδρία συμπίπτει με μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, η Σλοβακία σε αυτή την πρώτη της Προεδρία θέλει να προσφέρει νέα ενέργεια. Το Εθνικό Πρόγραμμα της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια αντανάκλαση της φιλοδεξίας να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της Ένωσης και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Το όραμα της Προεδρίας λοιπόν βασίζεται σε δύο πυλώνες. Πρώτον, μια θετική ατζέντα και δεύτερον, την εξέβρεση βιώσιμων λύσεων. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να υλοποιήσει έργα και προγράμματα που αποφέρουν πραγματικά ωφέλη στους πολίτες και την οικονομία. Στη διάρκεια της Προεδρίας θέλουμε να προωθήσουμε λύσεις που δεν απαντούν μόνο στις τρέχουσες εξελίξεις και προκλήσεις, αλλά λαμβάνουν ε, υπόψη τους και το μέλλον. Είμαστε αποφασισμένοι να δράσουμε με ειλικρίνεια όσον αφορά την ε, εκπλήρωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα λοιπόν έχω την ευκαιρία να σας ε, μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα, τα σλοβακικά, για τα θέματα της έρευνας, της επιστήμης και του διαστήματος. η κύρια φιλοδοξία λοιπόν της Σλοβαϊκής Προεδρίας στον τομέα της έρευνας, της επιστήμης και της, του διαστήματος είναι η ενίσχυση της, ε, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων της ε, Ένωσης. Στην ε, σημερινή δυναμική κοινωνία πρέπει να είμαστε προσανατολισμένοι στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και δυνατοτήτων. Εμείς πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη του κάθε πολίτη. Είτε μιλούμε για συμπεριφορά, είτε για δεξιότητες, το ταλέντο είναι πραγματικά ένας φορέας προώθησης της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης. Τις επόμενες ε, δεκαετίες η έρευνα και η καινοτομία θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως προς τη διατήρηση του ηγετικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Η Σλοβακία πιστεύει στη δύναμη των ιδεών και στη δυνατότητά τους όχι μόνο να ενισχύουν την ε, οικονομία αλλά και να βοηθούν στην εξέλιξη της ίδιας της κοινωνίας. Εμείς λοιπόν θα έχουμε μια προσέγγιση μέλλοντος στραφή προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία με ιδιαίτερη εστίαση στη νέα γενιά. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας επιδιώκουμε να θεσπίσουμε μέτρα για την ενίσχυση και την προαγωγή των νέων επιστημόνων, την ενίσχυση των ε, σταδιοδρομιών των νέων ανθρώπων στα πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε πώς από κοινού μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες και να άρουμε υπάρχοντα εμπόδια προκειμένου να οικοδομηθεί ένα ελκυστικό οικοσύστημα το οποίο θα επιτρέπει στους νέους επιστήμονες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους προκειμένου να διαχέουν και να αναπτύσσουν περαιτέρω καινοτόμες ιδέες. Από αυτή την άποψη η Σλοβαϊκή Προεδρία θα προσπαθήσει να ε, καταλήξει το Συμβούλιο σε συμπεράσματα προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα γενιά Ευρωπαίων ερευνητών με ενίσχυση της κινητικότητας και με ενίσχυση της ελκυστικότητας μιας ακαδημαϊκής καριέρας και προκειμένου να εμφυσίσει στους νέους επιστήμονες ένα ανοιχτό πνεύμα όσον αφορά την επιστημονική γνώση. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αυτά θα έχουν ως παράρτημά τους την διακήρυξη της Μπρατισλάβας που θα είναι ένα μανιφέστο νέων ερευνητών το οποίο έχει συνταχθεί από μια ομάδα εξαίρετων νέων επιστημόνων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από εμπλεκόμενους φορείς και ενώσεις και ομοσπονδίες που έχουν μεγάλη παράδοση στη συνεργασία με νέους ερευνητές. Η Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν καινοτομία και Έρευνας επίσης ε, συμμετέχει στη σύνταξη και τη διαμόρφωση του σχεδίου κειμένου. Έχουν ήδη γίνει πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις σε σχέση με αυτό το θέμα, συμπεριλαμβανομένου και του σεμιναρίου που έγινε στις 18 Μαρτίου στις Βρυξέλλες με εκπροσώπους των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας αλλά και με τη συμμετοχή νέων ερευνητών έπειτα, ε, η οποία μάλιστα, το οποίο ακολουθήθηκε από μία ε, επίσκεψη νέων Σλοβάκων επιστημόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες στις 30 Ιουνίου. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν μέχρι στιγμής κυρίως στους, ε, στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι επιστήμονες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τρόπους που μπορούν αυτά να ξεπεριαστούν. Τα αποτελέσματα και τα πορίσματα αυτών των συζητήσεων και διαβουλεύσεων αλλά και ε, των συζητήσεων που έγιναν μεταξύ των Υπουργών ε, έρευνας και κοινοτομίας στις 18 και 19 Μαΐου ε, ε, φετινού έτους θα συμπεριληφθούν και αυτά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε μορφή παραρτήματος και θα συζητηθούν και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας που θα διοργανωθεί στις 29 Νοεμβρίου φέτος. Μια άλλη προτεραιότητα θα είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου οικοσυστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ιδιαίτερη εστίαση στο πώς μπορούν να, να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους ερευνητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίως από τη σκοπιά των νεοπαγών εταιριών και των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν αναμφίβολα πρόσφορο έδαφος για τη διάχυση της έρευνας και της γνώσης. Σκοπός μας είναι να ε, ξεπεράσουμε νομικά και μη νομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν αυτού του είδους εταιρείε σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το οποίο έχει ως στόχο του να ενισχύσει και να προωθήσει τεχνολογίες εχμής όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αποκτήσει ηγετικό ρόλο, είναι ένα από τα εργαλεία που θα αξιοποιήσει η Σλοβακική Προεδρία προκειμένου να ενισχύσει την καινοτομία στον τομέα των επιχειρήσεων. Η διεύρυνση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 επίσης αποτελεί μια από τις μεγάλες προτεραιότητες της Προεδρίας μας. από την αναθεώρηση του προγράμματος πλαισίου 7 και την ενδιάμεση αναθεώρηση του ορίζοντα 2020 σκοπεύουμε να ε, διεξάγουμε συζητήσεις για τη μεγαλύτερη συμμετοχή και νέων φορέων στο πρόγραμμα αυτό. Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Ορίζοντας 2020, θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει και να προωθεί την αριστεία, στην καινοτομία και την έρευνα σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμη πολλές εξαιρετικές ερευνητικές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες ακόμη δεν, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 και αυτή η επέκταση, η διεύρυνση του προγράμματος θα μπορούσε να αναδείξει σημαντικές ευκαιρίες που προτείνει και που προσφέρει μάλλον το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Διάστημα και σχετικές υπηρεσίες, εφαρμογές και τεχνολογία. Όλα αυτά μπορούν να προσφέρουν ε, λύσεις σε υπάρχοντα αλλά και μελλοντικά προβλήματα. Η στατική για το διάστημα και η διαρρεύνηση του διαστήματο ε, είναι πολύ σημαντικό ο κλάδο μια ε, ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά, όπω είναι και η αυτοκινητοβιομηχανία, τεχνολογία και πολλοί άλλοι τομεί που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών μα. Επηρεάζουν ολόκληρο τον πληθυσμό λοιπόν. Ε, έχουμε επίγνωση των δυνατοτήτων ε, αυτής της ε, στρατηγικής και αυτής της ε, διαστημικής τεχνολογίας. Γι' αυτό και ορισμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ρωσία, έχουν τεθεί επικεφαλής αυτής της προσπάθειας και δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση. Θεωρούμε ότι και εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την οδό ε, θα βασιστούμε στις ε, εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ε, τεχνολογία και έτσι θα καταρτήσουμε την στρατηγική μας για το διάστημα, καθώς θα προσπαθήσουμε και εμείς να ηγηθούμε σε ένα τόσο στρατηγικό τομέα, σε μια υψηλά ανταγωνιστική αγορά. Είναι πολύ σημαντική από αυτήν τη σκοπιά η ετοιμότητά μας από πλευράς έρευνας, βιομηχανίας, υποδομών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να λειτουργήσουμε αυτά τα ε, προγράμματα. Η Προεδρία μας σκοπεύει να ε, παρακολουθήσει τι συμβαίνει με το θεματολόγιο για την συνεργασία νέου επίπεδου ε, για τις διαστημικές λειτουργίες. Θεωρούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει ε, τέτοιες συμφωνίες ε, για έναν ευρωπαϊκό διαστημικό χώρο μεταξύ κρατών μελών επιτροπής και ε, του αντίστοιχου ευρωπαϊκού φορέα. Υπάρχει συνεργασία και υπάρχει και πρόοδος, όμως είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την οδό, σε αυτό το διάλογο, προκειμένου να καταλήξουμε και να καταφέρουμε να πετύχουμε μία ε, κοινή συνεκτική και στρατηγική διαστημική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ε, θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε τους νέους επιστήμονες στη διαστημική έρευνα. Θέλουμε να προωθήσουμε λοιπόν αυτό το τομέα και τους επαγγελματίε του κλάδου, καθώς και τα συναφή επαγγέλματα του κλάδου. Ο Πρόεδρος μας θέλει να ε, θεσπίσει μια στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς φορείς και τον Ευρωπαϊκό Φορέα Διαστήματος ε, μέσα στα επόμενο διάστημα, ιδίως ότι αφορά τα προγράμματα Κοπέρνικος και Γαλιλαίος, που μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τους παρόχους, ε, τη βιομηχανία και την αγορά. Και τα δύο προγράμματα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ενεργούν ως ε, κινητήρι μοχλή ανάπτυξης και ερευνητικής προόδου το οποίο με τη σειρά του θα βοηθήσει και τη βιομηχανία και τις μικρές επιχειρήσεις. Η Προεδρία μας θέλει επίσης να ακολουθήσει το έργο της Ολλανδικής Προεδρίας σε ό,τι αφορά τη στενή συνεργασία με τον Κομισιόν, τα κράτη-μέλη και τον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Φορέα για την κατάρτιση και υλοποίηση μιας κοινή ευρωπαϊκής στρατηγικής για το διάστημα θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αναπτύξουμε ε, τις προτεραιότητές μας σε αυτούς τους τομείς ε, επιστήμης, έρευνας και διαστήματος, όχι μόνο στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, αλλά και σε άλλες τακτικές ή και ad hoc συνεδριάσεις που θα διοργανώσουμε και στις Βρυξέλλες και στη Σλοβακία. Κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα που θα γίνει 18 και 19 Ιουλίου στην Βρατισλάβα θα συζητηθεί ένα σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα στήριξη νέων ερευνητών, ε, ούτω ώστε να καταστήσουμε μια σταδιοδρομία στην, ε, στον ακαδημαϊκό κύκλο πιο ελκυστική και να ενισχύσουμε την, ε, τις επενδύσεις και στον τομέα αυτό. Θέλουμε επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ανάπτυξης και διαμόρφωσης ενός ε, ελκυστικού περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για καινοτόμες μικρότερες επιχειρήσεις. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ε, τις προϋποθέσεις για τους ερευνητές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην υπουργική διάσκευση της COST φέτος το Σεπτέμβριο θα εξετάσουμε τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας ε, στον στην επιστήμη και την τεχνολογία στο πλαίσιο της ε, σύνδεσης και συμφωνίας COST. Μαζί με την Επιτροπή θα διοργανώσουμε και μία συνεδρίαση ε, δικτύωσης ICT ε, που απευθύνεται βρέως στο κοινό και θέλει να ενημερώσει ε, το ευρύ κοινό λοιπόν για το πώς μπορεί κανείς να φτιάξει drafts για προτάσεις υπό τα πολύ γνωστά αυτά προγράμματα όπως το ορίζουν το 2020 και έτσι θα έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να διαμορφώσουμε ποιοτικέ ε, σχέσεις, ε, εταιρικέ σχέσεις στο χώρο της ακαδημίας, της βιομηχανίας, της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και στις μικρόμεσες επιχειρήσεις. Το θέμα της έρευνα και καινοτομία στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της Ενεργικής Ένωσης θα είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της διάσκεψης που ε, θα γίνει στα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, της CEEC. E e Διοργανώνεται συνήθως από την προεδρεύουσα χώρα και τη σχετική ε, διάσκεψη της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής. Θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε τα πιο συναφή ζητήματα που αφορούν την τρέχουσα ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, καθώς και την πολιτική μας και την έρευνα και κοινοτομία. Θέλουμε επίσης να εντοπίσουμε και νέες ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας. Ε, κατά τη αυτών των ημερών θα έχουμε και μια ειδική διοργάνωση για τις ανθρώπινες επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες ε, για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες προκλήσεις όπως είναι η ενεργία, η οικονομική ανάπτυξη, ε, κοινωνικές αλλαγές, μετανάστευση, ξενοφοβία και καταπολέμηση ξενοφοβίας πιο συγκεκριμένα. Μια διεθνής διάσκεψη για την επανακριβομηχάνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο 2016 θα διοργανωθεί επίση σχετικά με την νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, προηγμένα υλικά και ε, τεχνολογία παραγωγής. Σκοπός της οργάνωσης αυτής είναι να αναδείξει τον ρόλο της έρευνας ε, και τεχνολογίας και καινοτομίας ε, στη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και πιο συγκεκριμένα για την επανεκβιομηχάνηση της Ευρώπης. δίνοντας επαγγελματική στήριξη και καθοδήγηση για τους επιστήμονες. Αυτό θα είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που θα ασχολήσει ε, ένα ε, εργαστήρι που θα διοργανωθεί με τον όρο ε, «Σταδιοδρομία Παύλα Ερευνητή. Και στις 23 Νοεμβρίου θα έχουμε ένα ειδικό εργαστήρι για την καινοτομία, για τη στήριξη τη αριστεία στην έρευνα και καινοτομία και την διεύρυνση της συμμετοχή στο πρόγραμμα Horizon 2020. Επί ευκαιρία να σας ενημερώσω ότι το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα ω προ το τμήμα τη έρευνα, η Προσλοβική Προεδρία, θα γίνει στι 29 Νοεμβρίου 2016. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και ε, ελπίζω να συνεχίσουμε με τη συνεργασία μα και στο μέλλον. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την ομιλία σα σήμερα εδώ σχετικά με τι προτεραιότητε ε, τη Σλοβακική Προεδρία στον τομέα τη έρευνα και καινοτομία και στον ορίζοντα 2020. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση. Εξ ονόματο του Λαϊκού κόμματο, ο συνάδελφο Πίπερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την εντυπωσιακή αυτή παρουσίαση των προτεραιοτήτων σας στη διάρκεια της Προεδρίας σας. Δύο ερωτήματα έχω. Το ένα αφορά το θέμα της έρευνας. Εδώ με αναφερθήκατε στην οικολογική έρευνα και ότι θέλετε σε αυτήν να συμμετάσχουν ιδίω οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για έναν πολύ θετικό και σωστό στόχο. Ποια όμως θα είναι η σχέση αυτού του στόχου που θέτετε εσείς με το Ταμείο Juncker. Ποια θα ήταν η γνώμη σας δηλαδή ε, ποια είναι η γνώμη σας για το γεγονός ότι έχει εκφραστεί η πρόθεση να μεταφερθούν κονδύλια από την έρευνα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποια είναι η δική σας γνώμη. Ε, έχετε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα στη δική σας χώρα από αυτό το Ταμείο Ιούνκερ. Θέλω να ρωτήσω δηλαδή πώς συνδυάζεται η έρευνα με αυτό το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερο ερώτημα αφορά το διάστημα και τη σχετική στρατηγική. Όταν μιλούμε για ευρωπαϊκή πολιτική για το διάστημα, αυτό που εμένα μου λείπει πάντοτε είναι ποιο είναι το συγκεκριμένο όραμα. Δηλαδή, έχουμε το Γαλιλαίο, έχουμε και την Airbus και ίσως και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά όταν, όταν κανείς εξετάζει αυτήν την ευρωπαϊκή πολιτική για το διάστημα και λέει ότι θέλει να ασχοληθεί και να την ενισχύσει, να την προωθήσει, συγκεκριμένα πείτε μας, τι σκοπεύετε να κάνετε το επόμενο εξάμεινο και πώς μπορούν στην διαδικασία αυτή της ενίσχυσης της πολιτικής για το διάστημα να συμμετάσχουν οι μικρές μεσαίες επιχειρήσεις οι τοπικές κοινότητες. Ευχαριστώ. Η κυρία Λαβίτσκα έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας για να με καταλαβαίνετε. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που είχατε να μας πείτε. Ε, τα άκουσα προσεκτικά λοιπόν και έχω δύο ερωτήσεις. Σήμερα το πρωί συναντήσαμε εδώ τον, ε, ε, τον ε, Επίτροπο Αρμόδιο για Καινοτομία και Έρευνα και του έκανα λόγο για τις γεωγραφικές αποκλίσεις όσον αφορά ε, e, όσον αφορά τους δικαιούχους των προγραμμάτων για την έρευνα και την καινοτομία. Ε, και μάλιστα τον ρώτησα να μου πει αν έχει συγκεκριμένη ιδέα για την ε, αιτία αυτών των διαστάσεων και αν έχει κάποιο πρόγραμμα ε, να, και κάποιο τρόπο έτσι ώστε να αμβληθούν αυτές οι διαφορές. Ε, το ρωτώ και σε εσά αυτό. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει γίνει πολύ καλά αποδεκτό από τους πολίτες είναι το Erasmus Plus. Αλλά για τους νέους ε, ερευνητές, οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι πολύ ψηλές και επίσης ε, τα grants διαφέρουν από την μία χώρα στην άλλη. Και σε πολλές περιπτώσεις το επιτόκιο είναι πολύ μεγάλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ η πρόσβαση των νέων επιστημόνων ε, σε, αυτές τις, σε αυτά τα προγράμματα. Επανειλημμένα λοιπόν ρωτούμε και το ρωτώ και σε εσά αν προτίθεστε να αυξήσετε την χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στασενόφσκι θα πάρει τώρα το λόγο εξ ονόματος της ομάδας ECR. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή μας ασχολείται πολύ με την έρευνα, με την ε, τεχνολογία και με την ε, ε, βιομηχανία και την επιστήμη φυσικά. Το πρόγραμμά σας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος και σας συγχαίρω διότι ε, αναφερθήκατε στην ανταλλαγή ε, νέων ερευνητών και χαίρομαι γιατί βλέπω ότι το θέμα σας είναι ιδιαίτερος προσφυλές. Όλοι γνωρίζουμε ότι Πολλές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι γενικά, αλλά και οι νέοι επιστήμονες και ερευνητέ ειδικότερα. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα δύσκολο, να καταφέρει κανείς να βρει το δρόμο του όταν είναι νέος ερευνητής. Επίσης ξέρω ότι λόγω της περιπλοκότητας των δομών, λόγω ε, αυτού του πολύ βα, βαρέως οικοδομήματος γραφειοκρατίας, ξέρω ότι δεν θέλουν να ε, προσφεύγουν στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Προτιμούν να βρουν άλλο τρόπο χρηματοδότησης. Εγώ θα ήθελα να ανοίξετε κάπως τις πόρτες ε, στο, στα πλαίσια του ορίζοντα 2020. Πάντως, Πάντως, θα ήθελα να σας δω να ασχολείστε ιδιαίτερος με τους νέους επιστήμονες και τους νέους ερευνητές. Αναφερθήκατε επίσης ε, στην ε, έρευνα του διαστήματος, μεγάλα προγράμματα όπως ο Κοπέρνικος ή ο Γαλιλαίος. Που θα έχουν σημαντικότατες οικονομικές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία. Έχω ένα ερώτημα. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί κανείς να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τις ενημερώσει για την ύπαρξη του Γαλιλαίου και του Κοπέρνικου. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία ευαισθητοποίησης προκειμένου να χρησιμοποιούνται σε ευρύτερη κλίμακα τα προγράμματα αυτά και προκειμένου να καταστεί και σαφές στην κοινή γνώμη γιατί ακριβώς δαπανώνται τόσο μεγάλα ποσά σε αυτά τα προγράμματα. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα σταθούμε στο πλευρό σας, στην προσπάθειά σας να φέρετε ακόμη πιο κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη την επιστήμη και την έρευνα, γιατί σε τελική ανάλυση πρόκειται και για μία από τις σημαντικότερες συνεκτικές ουσίες του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. If Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ να απαντήσετε λοιπόν σε αυτές τις ερωτήσεις που σας υπέβαλαν οι συνάδελφοι. Επίσης ερωτήσεις ε, για το νέφος ε, computing και research. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα άλλο θα μπορούσε να είναι το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. Δηλαδή αυτή η νέα πρόταση. Ε, μάλιστα ο Επίτροπος ε, μας, που ήταν πριν ε, λίγο μαζί μας, ε, μας το παρουσίασε το πρωί. Και θα θέλαμε να ξέρουμε και την θέση σας, δηλαδή τη θέση της Σλοβακικής Προεδρίας. Στρέφαμε προς τους συναδέλφους, ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Α, κύριε Ρουμπίχ. Παρακαλώ, δεν σας είχα δει. Και υπέβαλα τα ερωτήματά μου εγώ. Ναι, συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο. Αλλά υπάρχει εκπρόσωπος Σλοβικής Προεδρίας και στην Επιτροπή Ανάπτυξης και είναι πραγματικά πολύ ε, ελπιδοφόρο το ότι βλέπουμε ότι η Σλοβακική Προεδρία θέτει προτεραιότητες που είναι σημαντικές για όλους μας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας. Ε, τι σκοπεύει να κάνει η Σλοβακική Προεδρία αν έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ και εγώ Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, είχα επισκέπτες, αλλά έκανα και εγώ δουλειά υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω και εγώ ένα ερώτημα, όσον αφορά το Γαλιλαίο και το Κοπέρνικο. Είναι δύο προγράμματα τα οποία μπαίνουν πλέον στην επιχειρησιακή, τη λειτουργική τους φάση και από αυτή την άποψη αυτό που θα δούμε το επόμενο διάστημα είναι η οικονομική αξιοποίηση αυτών των δύο προγραμμάτων. Τι σκοπεύετε να κάνετε. Πώς θα πείσετε τις εταιρείες να φύγουν από το GPS και να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τον Γαλιλαίο. Γιατί έχουν πραγματική καταβληθεί τε, τεράστιες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπόνηση αυτών των προγραμμάτων. Παρ' όλα αυτά, η ορατότητά τους είναι ελάχιστη στην κοινή γνώμη. Άρα, ε, νομίζω ότι σε εποχές όπως αυτή που διανύουμε σήμερα, αξίζει κανείς να αναδεικνύει και τα προγράμματα που έχουμε χρηματοδοτήσει και τα οποία έχουν στεφτεί με επιτυχία. Η κυρία Μπυρκόνεν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ αργοπόρησα λίγο, οπότε δεν άκουσα ολόκληρη την ε, παρέμβαση, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα στον κύριο Υπουργό διότι γνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση και η έρευνα ε, αποτελεί το θεμέλιο της ανάπτυξης ε, και της απασχόλησης. Πέρασα μας λοιπόν την άποψή σας για την εκπαίδευση και την έρευνα στην Ευρώπη Ποιες δηλαδή είναι οι ε, τομείς στους οποίους νομίζω ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες τώρα, ούτως ώστε να έχουμε καλής ποιότητας εκπαίδευση και έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και ανταγωνιστικότεροι μάλιστα στο μέλλον. Thank you for your question. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις Κύριε Υπουργέ, ε, εμείς από τη δική μας πλευρά υποβάλαμε τις ερωτήσεις που θέλαμε. Θα θέλαμε τώρα να ακούσουμε τις απαντήσεις σας και τα σχόλιά σας βεβαίως. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όσους έθεσαν ερωτήσεις Κάποιες ερωτήσεις μάλιστα συμπεριλάμβαναν και ορισμένες συστάσεις για τους επόμενους έξι μήνες, γιατί σε αυτές τις ερωτήσεις ε, κατάφερα και διέκραινα κάποιες πολύ θετικές ιδέες, τις οποίες και θα παρακολουθήσουμε στη διάρκεια της προεδρίας μας. Θα προσπαθήσω σε μία απάντηση να απαντήσω σε όλα αυτά τα θέματα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πολύ για την υποστήριξη που προσφέρετε στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο σχέδιο Juncker. Από αυτή την άποψη πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλές επιτυχημένες και νοτόμες ευρωπαϊκές εταιρείες και έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να σταθούν και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και βεβαίως έχετε δίκιο ε, είναι δικός μας στόχος να τις καταστήσουμε πιο ορατές αυτές τις εταιρείες. Να δώσουμε δηλαδή και τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη προκειμένου εκείνα να μας πούν τι ε, ε, είναι θετικό σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και ποια είναι τα εμπόδια και πώς θα μπορούσαμε να τα άρουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα ευνοεί την έρευνα με όφελος ε, μακροπρόθεσμο για τις μικρομεσαίε επιχειρήσεις. Τώρα, όσον αφορά τα, προγράμματα, ε, σαν αυτά που ανέφερε η κυρία Λαπίτσκα, το Μαρή Κιουρί, το τα κτλ, όλα αυτά τα προγράμματα είναι πολύ σημαντικά. Και αναγνωρίζω, καθώς ασχολούμαι με αυτά τα θέματα εδώ και πολλά χρόνια, ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία πρέπει να τα καταργήσουμε, να τα άρουμε τα οποία άλλωστε εμποδίζουν και την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. Και πολύ συχνά, πολλοί ερευνητέ δεν έχουν διάθεση να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του διοικητικού άχθους. Στην, στο Νοέμβριο θα γίνει αυτή η συνδιάσκεψη, αυτό το συνέδριο που σας ανέφερα, όπου νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις και να προσπαθήσουμε να ε, βρούμε και λύσεις, γιατί πραγματικά πρέπει να καταργήσουμε ορισμένα από αυτά τα εμπόδια που υπάρχουν και θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε και την συμμετοχή όλων των ε, μερών προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που χρηματοδοτούμε. Επίσης θα πρέπει να αποκαταστήσουμε και την ισορροπία μεταξύ νέων και παλαιών κρατών μελών. Άλλο ερώτημα. Ο κύριος Πίπερ και ο κύριος Τουχανόσκι αναφέρθηκαν στο ζήτημα του διαστήματος. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ερωτήσεις. Όσον αφορά την ομάδα εργασίας για το διάστημα, εμείς θα σας ε, κάνουμε και κάποιες παρουσιάσεις όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πράγματι χρησιμοποιούν διαστημικά δεδομένα. Και θέλουμε να δείξουμε στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το Κοπέρνικος έχει καταστεί ένα πολύ ελκυστικό πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια και είναι προφανές ότι πλέον είναι σχεδόν πλήρω λειτουργικό και έχετε δίκιο. Πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό το πρόγραμμα αυτό. Είναι λοιπόν ένας από τους στόχους που έχουμε θέσει το συγκεκριμένα, προκειμένου οι πολίτες μας να έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για αυτά τα προγράμματα, ώστε η κοινή γνώμη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μάθει περισσότερα πράγματα σε σχέση με τα συγκεκριμένα προγράμματα. Τώρα, να περάσω στο ερώτημα που αφορούσε το ευρωπαϊκό ερευνητικό υπολογιστικό νέφος. Ο δυναμισμός της ε, έρευνας βέως σημαίνει ότι η έρευνα διέρχεται από μια σειρά από αλλαγές. Χρειαζόμαστε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις γιατί βρισκόμαστε πλέον στον 21ο αιώνα και έχουμε πλέον τη δυνατότητα ταχείας επεξεργασίας μεγάλων όγκων δεδομένων. Και θα πρέπει και η ενιαία αγορά να ωφεληθεί από αυτές τις ε, νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Η Σλοβακική Προεδρία θα συζητήσει τα θέματα αυτά εντονότατα και η Κομισιόν θα παρουσιάσει και μια συγκεκριμένη στρατηγική για το πώς μπορούν να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ακόμη η κοινωνία. Ο ανοιχτός χαρακτήρας της επιστήμης είναι ένας τομέας που μπορεί να ωφελήσει και την έρευνα και την κοινή γνώμη, τους πολίτες, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Και ως αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι με αυτή τη νέα ανοιχτή προσέγγιση μπορεί να ωφεληθεί και η ίδια η έρευνα. Ρωτήσατε επίσης για την ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Κατά τη γνώμη μου, όλες οι νομικές πράξεις στα κράτη-μέλη, εκείνες που εστιάζουν στην ανώτατη εκπαίδευση, αναγνωρίζουν την σημασία της ερευνητικής δραστηριότητας Και βεβαίως όλες οι προσπάθειές μας πρέπει να κατατείνουν σε αυτό. Τη βελτίωση της ε, ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ψηλή ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βεβαίως συνδέεται άρρηκτα με την υψηλή ποιότητα της έρευνας. Και από αυτή την άποψη εμείς θα υποστηρίξουμε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ενίσχυση και τη βελτίωση της ποιότητας της έρευνας σε όλα τα επίπεδα άσκησης της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για τις απαντήσεις και τις παρατηρήσεις σας. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα να συζητούμε τόσο σημαντικά θέματα μαζί σας, όπως είναι η έρευνα, η καινοτομία, η παιδεία. Τώρα, κατά την έναρξη της ε, Προεδρίας σας, σας ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία στο έργο σας, γιατί η δική σας επιτυχία θα είναι μια επιτυχία ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που παρευρεθήκατε εδώ σήμερα μαζί μας που βρεθήκατε σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Uh, uh, Συνάδελφοι, πάμε στο θέμα 13. Μέτρα για την εξασφάλιση της, ε, για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Θα ήθελα να πω, κατά την έναρξη της αυτού του θέματος, κάποιες παρατηρήσεις. Ως εισηγητής επί του συγκεκριμένου προτινόμενου κανονισμού. Πρώτα απ' όλα, εκτός από τις 125 τροπολογίες που έλαβα για αυτό το σχέδιο έκθεσης, τα μέλη της Επιτροπής υπέβαλαν και άλλες 763 τροπολογίες, κάνοντάς τις συνολικά 888. Οι τροπολογίες αυτές αφορούν όλα τα σημαντικά θέματα της ε, πρότασης Κομισιόν, όπως είναι ο ορισμός του προστατευόμενου πελάτη, αλλά και των κοινωνικών ε, υπηρεσιών την αξιολόγηση κινδύνου, τις, τα σχέδια δράσης ε, πρόληψης, σχέδια έκτακτης ανάγκης και είναι επίσης πολύ σημαντικό. υποχρεώσεις των εταιριών φυσικού αερίου και την υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση κρίσης. Πολλές τροπολογίες επίσης αντικατροπτρίζουν και τη δική μου πρόταση να συσταθούν διάδρομοι εφοδιασμού έκτακτης ανάγκης. Πολλές τροπολογίες επίσης ζητούν την ενίσχυση των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ως μέτρο εξασφάλισης του εφοδιασμού με αέριο. So I should να ξεκινήσω από την αρχή. Είναι γενικές οι παρατηρήσεις που κάνω τώρα. Ο κανονισμός αφορά το πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλιστούμε σε περίπτωση μεγάλης μίζωνος κρίσης. Καταρχάς, εμείς πιστεύουμε στην ενιαία αγορά ενέργειας και στο βαθμό του δυνατού θα πρέπει να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες που προσφέρει η αγορά. Αλλά στις μείζονες κρίσεις χρειαζόμαστε αξιολογήσεις κινδύνου, χρειαζόμαστε προληπτική δράση και αντίστοιχα σχέδια δράσης, αλλά και σχέδια δράσης έκτακτης ανάγκης. Και ως έσχατο μέτρο Βεβαίως ελπίζουμε κάτι τέτοιο να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σχέδιο αλληλεγγύη. Δηλαδή μιλούμε εδώ για την αλληλεγγύη ως νομική υποχρέωση, ως έσχατο μέτρο πάντα, έτσι. Τι θα απαιτηθεί για να ορίσουμε τους προστατευόμενους πελάτες νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε μεγάλες δυσκολίες. Θα πρέπει να είναι ελάχιστος ο αριθμός προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ όλων των κρατών μελών και όλων των ευρωβουλευτών. Όμως, η μέθοδος αποζημίωσης είναι ένα θέμα που δεν είναι τόσο εύκολο να καταλήξουμε σε απόφαση. Θα είναι το πρώτο και πλέον δύσκολο θέμα που θα συζητήσουμε στο έργο μας με τους σκιώδεις εισηγητές. Δεύτερο θέμα. Περιφέρειες. Και πώς οι περιφέρειες θα πρέπει να λειτουργούν. αλλά και πώς θα παρουσιάζουν αξιολογήσεις κινδύνου, ε, σχέδια προληπτικής δράσης, σχέδια της ανάγκης, μαζί και με ειδικού διαδρόμους εφοδιασμού έκτακτης ανάγκης, που το οποίο θα μπορούσε να είναι κρίσιμη σημασία στο μέλλον. Και βρισκόμαστε σε επαφή με τους ε, παρόχους υπηρεσιών σε αυτόν τον τομέα. Και ένα τελευταίο πολύ σημαντικό στοιχείο αφορά την κοινοποίηση των ε, πιο σημαντικών συμβάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ των υστέρων. Ε, κοινοποίηση, όπως ξέρουμε, στην περίπτωση διακυβερνητικών συμφωνιών, ε, και συμβάσεων, εκεί αναμένεται κοινοποίηση εξάντε. Όμως στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση μιλούμε για εκ των υστέρων κοινοποίηση ορισμένων από τις πλέον σημαντικές τέτοιες συμβάσεις. Με τα θέματα ενεργειακής απόδοσης, τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν σε δύσκολες ε, περιστάσεις. Για μένα αυτό είναι σαφές. Ε, δεν θα ήταν κάτι πολύ δύσκολο να προσθέσουμε κάτι τέτοιο στην πρότασή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο τώρα στους Χιόδης. Εξ των Σοσιαλιστών, η κυρία Γκρίφιν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτον να σας ευχαριστήσω θερμά, Τζέρση, για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα για αυτό το φάκελο. Η ασφάλεια φωτιασμού φυσικού αερίου δεν μπορεί να επιτευχθεί ε, από ένα κράτος μέλος μεμονωμένα. Πρέπει να, να είναι αποτέλεσμα μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας. Εμείς θέλουμε με τις ε, τροπολογίες μας να στηρίξουμε την πρότασή σας για την βιωσιμότητα. Τονίζουμε το ρόλο της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης των ΑΠΕ, ε, καθώς και την ε, ενίσχυση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και τη μείωση ε, των εισαγωγών. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε τέτοια πολιτική μας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα περιβαλλοντικά και τα ζητήματα του κλίματος. Επομένως, θα πρέπει να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση και να μειώσουμε την κατανάλωση. Επίση, νέε υποδομέ φυσικού αερίου θα πρέπει να αντιποκριθούν μόνο σε πραγματική ζήτηση φυσικού αερίου ε, για να μην υπάρξουν χαμένε επενδύσει. Τέλο, πρέπει να αξιολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ε, παρόχου τρίτων χωρών ε, με βάση την βιωσιμότητά του θέλουμε μία ενοποιημένη προσέγγιση και για το φυσικό αέριο και για την ηλεκτρική ενέργεια. Στηρίζουμε την ιδέα της περιφερειακής συνεργασίας με ειδικούς διαδρόμους έκτακτες ανάγκης για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες κρίσεις. Ο διασυνοριακός και υπερεθνικός ε, τέτοιος κίνδυνος απαιτούν ενισχυμένη συνεργασία με πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ανταποκριθούμε σε πιθανές κρίσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, μέτρα ε, τα οποία θα υιοθετούνται από κοινού τα κρατη για τη ε, διαμόρφωση προληπτικών σχεδίων. Όμως τα περιφερειακά προγράμματα δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν τα εθνικά προγράμματα, τα οποία θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα. Συντονισμός λοιπόν όταν θα έχουμε εντοπίσει μείζονες κινδύνους. Προτείνεται λοιπόν αυτό το επίπεδο συνεργασίας από εσάς μέσω των ε, διαδρόμων εφοδιασμού έκτακτη ανάγκη και εμεί στηρίζουμε αυτή την πρότασή σα. Πρέπει να διευκρινίσουμε γενικά ότι αυτές οι περιφέρειες δεν αποτρέπουν από κανένα κράτο μέλο να συνεργάζεται με γειτονικέ χώρε πέραν της περιφερειάς τους. Και ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι μαζί σα μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ταρέζα, για τα σχόλιά σου. Επόμενο χειώδη εξ ονόματο του ECR, ο κύριο Τσέσα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και σας προσωπικά Διατρέξατε ήδη κάποια από τα σχόλια στις τροπολογίες γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και βεβαίως θα πρέπει ο καθένας να υποβάλλει τις δικές του απόψεις. Γνωρίζουμε ότι το σχέδιο έκθεσης καλύπτει ε, πολλές σημαντικές πτυχές της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου και βέβαια πρέπει όλο αυτό το ζήτημα να το εντάξουμε και στο πλαίσιο του προγράμματος Nord Stream 2 το οποίο αξιοποιείται και ως ένα γεωπολιτικό εργαλείο για το μέλλον. Κατά τη γνώμη μου, προφανώς αν εξετάσουμε την έκθεση και την προσέγγιση του εισηγητή, θα πρέπει να εξετάσουμε τον ρόλο που μπορούν να διαματήσουν οι περιφέρειες σε τυχόν ε, διακοπές ή προβλήματα το, της ε, ασφάλισης εφοδιασμού ό,τι αφορά την ε, ε, τυποποίηση, τη διαμόρφωση προτύπων, την ενίσχυση αλληλεγγύη και ούτω καθεξής για να αποφύγουμε τέτοιε ε, περιπτώσει έκτακτη ανάγκη. Πρέπει επίση να δούμε τι συμβαίνει με τι μακροπρόθεσμε εμπορικέ συμφωνίε που υπογράφονται μεταξύ επιμέρου παρόχων. Αυτή είναι η πρώτη μας ε, συζήτηση για αυτή την έκθεση. Και βεβαίως, αν εξετάσει κανείς το αρχικό έγγραφο, Νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω με τη θέση του εισηγητή ότι μέχρι τώρα ως προς τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών σε αυτό το πεδίο είναι ελλειπή θα έλεγα. Και εγώ έχω υποβάλει ορισμένε τροπολογίε και νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με τη διαμόρφωση αυτών των περιφερειών που προτείνει ο εισηγητής. Έχουμε το Acer, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, αλλά και, την και ο Ευρωπαϊκός νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να ενισχύσει αυτές τις ε, διατάξεις ως προς την ε, αντίστροφη ροή σε περιπτώσεις ε, κρίσεων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να δούμε τι συμβαίνει με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, και με τους επιμέρους ε, TSOs και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύονται όλοι οι πάροχοι ηλεκτρικής, ε, συγγνώμη, φυσικού αερίου, ανεξαρτήτως μεγέθους. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό στην έκθεση. Θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις ε, συμβάσεις φυσικού αερίου και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εξετάσουμε και να αναλύσουμε αυτές τις συμβάσει μεταξύ των παρόχων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, παρόχων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα εξετάσουμε στην έκθεση, αλλά εντάξει, όλα αυτά θα τα δούμε και στο μέλλον. Κλείνοντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Γιατί έχει ήδη ορίσει τι ημερομηνίε για τι ομάδε εργασία και μα έχει δώσει μια πολύ σαφή εικόνα για τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής εξ ονόματο της Γκούι, ο κύριος Μπενίτος Τιλουάγκα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι μόλις μου ήρθε ε, αυτό, αυτή η ε, βεντάλια που λέει ότι gas is not cool. Ε, αυτό βεβαίως καταδεικνύει ότι όλοι οι πολίτες παρακολουθούν από κοντά το θέμα αυτό. Μια και μιλάμε για την προμήθεια του φυσικού ε, αερίου, πρέπει να σας πω ότι έχουν υπάρξει διαρροές ε, τώρα τελευταία ε, και αναφέρονται σε μια δεσμευτική νομικά συμφωνία όσον αφορά περιορισμούς του φυσικού αερίου που μπαίνει στο εμπόριο. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγουν οι πόρτες για την περαιτέρω εισαγωγή ορυκτών καυσίμων, δηλαδή συγκεκριμένα έρονται οι περιορισμοί για τις ε, ε, εισαγωγές ε, από τις Ηνωμένε Πολιτείε δεν βγαίνουν δε από αυτές τις εισαγωγές οι παραγωγέ οι οποίε έχουν προκύψει από υδρορογμάτωση. Αυτό βεβαίω καταλαβαίνετε ότι αντιτίθεται ε, πλήρως ε, στη Συμφωνία των Παρισίων. Εμεί ε, γι' αυτό και για άλλου λόγους, αλλά και γι' αυτό δεν συμφωνούμε με την Συμφωνία TTIP και γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι ήδη υπάρχουσες υποδομές. Πριν δημιουργήσουμε καινούριε υποδομέ θα πρέπει να δούμε και τις υφιστάμενες δυνατότητες αλλά και την ε, δυνατότητα ενδογενούς ε, παραγωγής ενέργειας μέσα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς επίσης και αποτελεσματικότερη χρήση όλων των εργαλείων που έχουμε τώρα. Any other request for floor? Ε, ζητά κάποιος άλλος τον λόγο από τη συνάδελφη. Δεν βλέπω. Α, κύριε Ταμπουράνο. Ναι, παρακαλώ, δεν σας Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Μπουζέ και ευχαριστώ πολύ και για την καλή συνεργασία που είχαμε ε, στη διάρκεια της προετοιμασίας. Εμείς ε, συμφωνούμε με ορισμένα τμήματα της πρότασης Μπουζέ και κυρίως δε με το θέμα των διασυνοριακών διασυνδέσεων ε, και βεβαίως ε, λέμε ότι στις διαμεθοριακές συνδέσεις θα πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουμε όλο το δυναμικό. Μας εκπλήσει που δεν έχει ληφθεί υπόψη συστηματικά το θέμα της αντίστροφης ε, ροής. Δυστυχώς όμως έχουμε κάποιες περιπλοκές όσον αφορά την σύσταση των περιφερειών. Αυτή η περιφερειοποίηση μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Ε, θα μπορούσε λύση να αφορά μια ενδεχόμενη ε, ευελιξία όσον αφορά εθελούσιες περιφερειοποίησης. έτσι όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα 1. Αυτό που μας προβληματίζει αρκετά πάντως είναι το γεγονός ότι δεν θα θέλαμε ο κανονισμός αυτός, ο οποίος αφορά ε, στην ασφάλεια, ε, να μην ε, αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο το δούριο ύπο για τη δημιουργία νέων υποδομών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλές υποδομές οι οποίες σαφώς υπολειτουργούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε τη στιγμή που συμβαίνει αυτό να δημιουργηθούν, να χτιστούν κι άλλες. Ούτε θέλουμε να χτιστούν επιπλέον ε, αγωγοί οι οποίοι ε, στην ουσία θα αντλήσουν χρηματοδότηση ε, από την από, την ενεργειακή, από τα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης. Επίσης μας προβληματίζει πάρα πολύ η διαρροή ε, του ε, TTIP, ε, η οποία είναι διαρροή την οποία οφείλουμε στην ε, Greenpeace της Γερμανίας. Μας απασχολεί πολύ γιατί στην ουσία ε, επιματέω οδηγείται όλη η δουλειά που έχουμε κάνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αλλού βέβαια. Αυτό το, αυτή η διαρροή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρότατα υπόψη. Επίσης, δύο τελικές σκέψεις έτσι ευρύτερης εμβέλειας. Ε, το θέμα του Λουκίν καθώς επίσης ε, και οι ενεργειακές πολιτικές ε, να, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στον κόσμο, ειδικά δε σε αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, οι νόμοι της φύσης είναι αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν. Βεβαίως θα μου πείτε και τον νόμο της βαρύτητας τον έχουμε και νικήσει τη στιγμή που μπορούμε και πετάμε με το αεροπλάνο, αλλά κάποια στιγμή οφείλουμε να προσγειωθούμε. Α, κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να σκεφτούμε ε, όσον αφορά την χρήση των ορυκτών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να λειτουργήσουμε ε, με τρόπο ώστε να μην δημιουργηθούν φαινόμενα lock-in. Έχω και άλλα βέβαια να σας πω πολλά, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα, δεν έχουμε και το χρόνο. Uh, Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε για αυτές τις παρατηρήσεις. Ο κύριος Σον Κέλλη. Ευχαριστώ. Το ζήτημα της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο είναι πολύ σημαντικό και έχουμε εξετάσει το θέμα αυτό υπό το φως ε, και της απόφασης COP21 όπως έχει συζητηθεί εδώ πολλές φορές. Ταυτόχρονα το φυσικό αέριο είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον ορυκτό καύσιμο, καύσιμο και θα χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια ακόμη. Άρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ασφάλεια εφοδιασμού στην Ευρώπη. Επίσης βεβαίως είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε τις οδούς προμήθειας και εφοδιασμού και από αυτή την άποψη είναι σημαντικό να εξετάσουμε και το ζήτημα του LNG. Στη δική μου χώρα, έπειτα από το Brexit, εμείς θα βρεθούμε σε ιδιαίτερη και δύσκολη θέση. Γιατί εμείς συνδεόμαστε μέσω ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Άρα, σε 5-10 χρόνια θα εξαρτώμαστε απόλυτα από το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο μάλιστα δεν θα είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να υπάρξει μια διαφοροποίηση των ε, οδών προμήθειας. Και δεν καταλαβαίνω όλη αυτή τη φιλολογία κατά του TTIP. Όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δώσει την έγκρισή τους για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Και δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή αν είμαστε κατά ή υπέρ, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα τι έχουν, ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης. Επίσης, ανησυχώ λίγο με το να δίνεται ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στις διαρροές της Greenpeace και άλλων. Με, με διαρροές δεν γίνεται πολιτική. Ούτε πιστεύω ότι ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι πρέπει εμείς να καθόμαστε και να βασιζόμαστε σε διαρροές. Εμείς λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουμε την εντολή που μας έχει δοθεί να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας. Έτσι θα σημειώσουμε πρόοδο και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι από τη δική μας κοπιά θα παρέχουμε κάθε υποστήριξη προς εσένα προκειμένου να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση για το θέμα του, της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Στέφαν Μόζελ από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, από τα, πιο, από τα πλέον αξιόπιστα μέλη της ε, υπαλλήλου μάλλον της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ, ευχαριστώ και του ευρωβουλευτές για την πρόσκληση αλλά και για το γεγονός ότι μας δίνεται η δυνατότητα να συζητούμε διάφορα θέματα σε διάφορες περιστάσεις. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό το θέμα που συζητούμε είναι ένα νέο θέμα στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης Μιλούμε πάντοτε για την ενεργειακή αποδοτικότητα, για τον μετριασμό της ζήτησης, την βιωσιμότητα, το κλίμα και πιο συγκεκριμένα έχουμε την επιτυχία του COP21 και στο πλαίσιο αυτό ανακύπτει το ερώτημα ποιος θα είναι ο ρόλος του φυσικού αερίου. Κατά τη γνώμη μας το φυσικό αέριο θα είναι μια σημαντικότατη support uh, renewables um, um, energy efficiency will have to forward θα είναι μια σημαντικότατη πρόοδος που θα μπορέσουμε να σημειώσουμε ε, Ωστόσο η ζήτηση δεν θα μειωθεί τόσο ώστε να μπορούμε να απεμπλακούμε πλήρως από τις αγωγέ. Οι αγωγέ θα υπάρχουν και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε στη διάθεσή μα τους πόρου που χρειαζόμαστε και πρέπει να αποφύγουμε, όπω είπαν και άλλα μέλη της ε, την, ε, τις υπερβολικές ε, επενδύσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, πραγματοποιηθούν εκείνες οι επενδύσεις που είναι πραγματικά αναγκαίες και να διασυνδεθούν οι υπάρχουσες υποδομές προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση στους πόρους φυσικού αερίου για να αποφεύγονται τυχόν διακοπές εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό φυσικά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παγιδευτούμε στη χρήση του άνθρακα. Άρα καλύτερα να μην γίνουν μεγάλες απαντήσεις, αλλά καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών, έτσι θα τα καταφέρουμε. Θα κάνουμε ένα άλμα λοιπόν προς τα εμπρός, ε, με αυτή την ε, οδό ε, που σας παρουσίασα. Το είπε και ο κύριος Μπούζεκ στην εισαγωγική του ομιλία. Εμείς Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την προσέγγιση του Κοινοβουλίου. Διάδρομη προμήθειας ε, εφοδιασμού μάλλον έκτακτης ανάγκης. Ανάλυση εκ των προτέρων. Συγκέντρωση όλης της εμπειρογνωμοσύνης με επικεφαλή την Έντσο. αξιολογήσει κινδύνου και ανάπτυξη περιφερειακών σχεδίων θα χρειαστούν βεβαίως και εθνικά στοιχεία, εθνική συμβολή και στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική και σε βάθος συζήτηση σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου κανείς να μην πληγεί από τα μέτρα που θα ληφθούν. Και βεβαίως θα πρέπει να θυσπιστούν και διασυνοριακά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτή η πραγματική συνεργασία, η διαπεριφερειακή. Η αλληλεγγύη, όπως είπε και ο κύριος Μπούζεκ, είναι ένα έσχατο μέτρο, αλλά αποτελεί και μια συμβολική αντανάκλαση, αντανάκλαση μιας πραγματικής ενεργειακής ένωσης και γι' αυτό ως μηχανισμός εξασφάλισης θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι πρακτικές διευθετήσεις θα είναι λειτουργικές το Σεπτέμβριο θα γίνει και μια σχετική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να αποσαφινιστεί και το τι ακριβώς θα χρειαστεί στην, στο μέλλον και τι ακριβώς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει η νομοθετική πρόταση αλλά και οι κατευθυντήρες γραμμές της ε, Κομισιόν. Στις συμβάσεις χρειάζεται να βρούμε μια ισορροπία ανάλογα, ε, ανάμεσα στο τι χρειάζεται τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν όσον αφορά τους περιορισμούς διατηρώντας ταυτόχρονα το διοικητικό άχθος όσο το δυνατόν χαμηλότερα, θα πρέπει να υπάρξει και μια εκ των υστέρων αξιολόγηση της όλης διαδικασίας και βάσει αυτής θα θεσπιστούν και ορισμένες ρήτρες αποκλεισμού. Η Ενεργειακή Ένωση για εμάς αποτελεί την φυσική συνέχεια των προσπαθειών για την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού. Θέλουμε τη συνεργασία με την Ουκρανία, τη Μολδαβία, την Λευκορωσία και είναι αμοιβαία επωφελής αυτή η συνεργασία στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης μέσω της, γιατί μέσω αυτής μειώνονται τα κόστη και αυξάνεται η αποδοτικότητα των ε, του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Υπάρχουν και ζητήματα όπως είναι ο προστατευμένος καταναλώτης, πελάτης, η βιωσιμότητα, οι ερευνητικέ επιπτώσεις από τις διαρροές φυσικού αερίου, LNG, και αποθεματοποίηση του φυσικού αερίου. Σε αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να έρθουμε σε στενή διαβόλευση με τις επιχειρήσεις, με τις εταιρείε. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να εξαταστούν και αλλού, σε άλλα βήματα και να συζητηθούν σε βάθος. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν που μας προσκαλέσατε εδώ και εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι σας. Ε, ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή συνεργασία. Νομίζω ότι συνεννοούμαστε αρκετά εύκολα. Ενδεχομένως να διαφωνούμε σε ορισμένα σημεία, όμως το πιο σημαντικό είναι να τα συζητούμε πολύ ανοιχτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τερέζα, αυτό που επεσήμανες για τους διαδρόμους έκτακτη ανάγκης, ότι αυτό μπορεί δηλαδή να λύσει ορισμένα ερωτήματα, να δώσει απαντήσεις και στη συνεργασία μεταξύ περιφερειών. Το ίδιο είναι η απάντηση και για τον κύριο Ταμπουράνο. Ζητήσατε ευελιξία. Αν επιπροσθέτως, όχι ως βασική λύση, αλλά συμπληρωματικά προσθέσουμε και τους ε, διαδρόμους της ανάγκης στις περιφερειές μας, θα δώσει κάποια ευελιξία. θα εντοπίζεται από τους ευρωπαϊκούς ε, TSOs και θα γίνονται αποδεκτοί από ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στην NSOG είναι έτοιμοι, είναι διατεθειμένοι να μας στηρίξουν, εκπροσωπούν 28 κράτη-μέλη. Είναι έτοιμοι λοιπόν όλοι αυτοί οι φορείς να συνεργαστούν μεταξύ τους και όχι να κατασκευάσουν ενδεχομένω, αλλά να εντοπίσουν διαδρόμους έκτακτη ανάγκης. Όπως ανέφερε ο Σον προηγουμένως, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα. Γιατί μία από τις ε, περιφέρειές μας ε, ενδέχεται να εξαφανιστεί. Δεν πρόκειται για επίσημο αίτημα της ε, Βρετανικής κυβέρνησης ακόμα. Ακόμα λοιπόν υπάρχει η περιφέρεια αυτή. Αλλά χωρίς ε, τη Μεγάλη Βρετανία θα τεθεί το ζήτημα στο μέλλον σίγουρα. Και επισημάνατε πολύ σημαντικά ερωτήματα όντω. Μετά, και αυτό που είπε ο κύριο Τσέσακ, αν κοινοποιούνται όλες οι συμβάσεις. Έχουμε χιλιάδες τέτοιε συμβάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιε από αυτές πραγματικά δεν είναι κρίσιμη σημασία για την ασφαλειά μας. Ας περιοριστούμε λοιπόν στις πλέον σημαντικέ από πλευράς ε, ασφάλεια εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν χρειάζεται να πάμε σε τέτοιο επίπεδο λεπτομεριών. Μπορεί να διαφωνήσουμε σε αυτό, εντάξει, αλλά όλα αυτά είναι μπροστά μας, θα τα συζητήσουμε. Σας καλό να τα σκεφτείτε πολύ καλά και με ψυχραιμία τις επόμενες εβδομάδες κατά τη διάρκεια των δικοπών σας. και να χρησιμοποιήσετε το φυσικό αέριο όπου θέλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Θα είναι πολύ σημαντική ε, έκθεση στην οποία θα βασίζονται και οι καταναλωτές μας, αλλά και για τις ενεργειακές επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τον κλάδο, τον ενεργειακό. Πρέπει πάντα λοιπόν να τους θυμόμαστε τους εκπροσώπους του ενεργειακού κλάδου, αν θέλουμε να προστατεύσουμε και τους καταναλωτές μας. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για την πολύ καλή συζήτηση. Θα συνεχιστεί η πολύ καλή αυτή προσπάθεια και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Τώρα θα περάσουμε στο σημείο 14 της μέσης διάταξης τελευταίο αλλά και εξίσου σημαντικό πριν τις διακοπές. Τα διάφορα θα είναι το τελευταίο τέλο πάντων, εντάξει αυτό είναι το πρώτο τελευταίο. Για το ETS, ε, μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ε, εισηγητής Φέντερικ Φέντερλεϊ. συντάχθηκε η γνωμοδότηση με βάση τον κανόνα 54 με επιμερισμένη αρμοδιότητα για ε, τις διαρροές άνθρακα μεταξύ άλλων. Πολλές τροπολογίες, 47 κατέθεσε ο εισηγητής. Για την Επιτροπή Ήτρε δεν είναι καθήλυν αρμόδια Παρ' όλα αυτά, είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η έκθεση. Επομένω και η συζήτησή μα ε, μπορεί να είναι ε, πολύ σημαντική για μια ανταγωνιστική βιομηχανία, αλλά και για του περιβαλλοντικού μα ε, στόχου. Συνάδελφε κοιτά. παρακαλώ Φρέντερικ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για αυτό το σημαντικό φάκελο με τα είδαμε ότι υπάρχει μια ισχυρότερη θέση της ΙΤΡΕ χάρη στις προσπάθειες του Προέδρου Μπουσέκ. Για ορισμένα τμήματα του ETS έχουμε την ίδια θέση με την Επιτροπή ΕΜΒΗ, το οποίο είναι σημαντικό για την Επιτροπή μας. Γι' αυτό και στην έκθεση έχουμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση ε, στη δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά θα εκφέρουμε γνώμη για όλα τα τμήματα του ETS. Πρώτον, Επί της διαδικασίας υπήρξε μια συζήτηση ε, με βάση την έκθεση στην Επιτροπή Ήτρε. 780 τροπολογίες ε, έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι του Κοινοβουλίου και θα εξετάσω πολλές από αυτές ε, και θα δούμε ποια μηνύματα μπορούμε να συνεγάγουμε από όλα αυτά. Με οικονομικό αποδοτικό τρόπο λοιπόν οι περικοπέ των εκπομπών εξουδίων τα άνθρακα, για τη διαρροή του άνθρακα και πώ θα βασιστούμε στη Συμφωνία των Περισσίων, τα βασικά ζητήματα. Για τη διαρροή εξουδίων του άνθρακα έχουμε μια στοχευμένη προσέγγιση όπω πρότεινα στην έκθεσή μου, αλλά θέλουμε επίση να εξετάσουμε και την πρόταση τη Κομισιόν με έναν ε, τέτοιο δεσμευτικό κατάλογο. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, αλλά και εγώ και οι Σκιώδης καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να υπάρχει πλειοψηφία για την έκθεση στην Ήτρε. Αυτό σημαίνει ότι όλοι τελικά θα πρέπει κάποιους συμβασμούς να κάνουμε. Για, με βάση τα στοιχεία ε, υπάρχει μεγάλη στήριξη για το δεύτερο ζήτημα. Για τα benchmarks υπάρχουν ορισμένες διαφορές. ανάλογα με το αν θέλουμε προσέγγιση νέων δεδομένων ή ε, flat rate που προτείνει η Κομισιόν. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να περάσουμε σε πλήρη συλλογή δεδομένων, ίσως έτσι ε, να τιμωρήσουμε αυτούς που κινήθηκαν γρήγορα και ήδη από τώρα, σε πρώιμη φάση, έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις και διερευνούν τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή για να ε, μειώσουμε τις εκπομπές. Ίσως θα ήταν ε, πιο ωφέλιμο σε όσους δεν έχουν κάνει ακόμα κάποια κίνηση. Μάλλον τελικά θα καταλήξουμε σε συμβιβασμό μεταξύ των επιμέρους απόψεων. Για την αποζημίωση του κόστους υπάρχουν τροπολογίες προς πάσα κατεύθυνση. Ορισμένοι βουλευτές θέλουν ε, εθελούς αποζημίωση, άλλοι θέλουν καμία αποζημίωση. Άλλοι θέλουν υποχρεωτική αποζημίωση με βάση τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και θέσπιση καθεστώτος αποζημίωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα είναι δύσκολο να λυθεί αυτό το ζήτημα, αλλά σίγουρα θα καταφέρουμε κάτι να κάνουμε. Για να εξεύρουμε ένα συμβιβασμό προς την μη κινητοποίηση του ε, διακλαδικού συντελεστή διόρθωση και αυτό θα είναι πρόβλημα. Όμως ακούω από τους συναδέλφου ότι αυτό είναι ο βασικός στόχος. Σε όσου έχουμε υποσχεθεί ε, δωρεάν ποσά να τα πάρουν. Κάποιοι έχουν ακούσει ακόμη και 20%. Προς το παρόν θα τους αφαιρεθεί λόγω του συντελεστή διόρθωσης. Ε, Πώ θα ηγηθούμε της ε, καινοτομία. Πολλοί συνάδελφοι λένε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερο και πιο ισχυρό ταμείο καινοτομία, προκειμένου να είναι πραγματικά σημαντικό εργαλείο για την κλιμάκωση αυτών των προσπαθειών. Για την πηγή ε, είναι, οι απόψεις διήστανται. Έχουμε δύο ουσιαστικά κατευθύνσεις σε όλες τι τροπολογίες υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα επιμέρου ταμεία και κατά πόσο θα πρέπει τα όρια να δίνονται από ε, το μερίδιο δημοπρασιών ή από τις ελεύθερες ε, ποσότητες που κατανέμονται. Ε, ενοποίηση της αγοράς ενέργειας, ε, ιδίως ό,τι αφορά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ε, στα κράτη-μέλη χαμηλών εισοδημάτων. Υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, αυτό είναι θετικό με βάση και του μακροπρόθεσμου ε, περιβαλλοντικού στόχου τη Ένωση. Όμω υπάρχουν πολλέ τροπολογίε που κινούνται στην την αντίθετη κατεύθυνση. Η διακυβέρνηση για την καθοδήγηση στη χρήση των ταμείων είναι κρίσιμη σημασία για να μην υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρική ενέργεια των σύγκρατων μελών. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει αντίθετα προς την εργασία η οποία καταβάλλεται για την επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης. Επίσης, ε, συμφωνώ να μην υπάρχει καμία αρνητική ε, διάδραση με το EUTES. Τελευταίο στοιχείο, ευρία ε, συνένεση όσον αφορά το σύστημα ε, των, ε, της ανταλλαγής και εμπορίας εκπομπών και τις αποφάσεις του Παρισιού. Μετά από τη διάσκεψη του Παρισιού έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη συνθήκη των Παρισίων για να δουν οι διάφορες χώρες τι πρέπει να επικαιροποιηθεί και τι να διευρυνθεί εισαχθεί ε, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν κατά αυτή την έννοια να γίνουν οι σωστοί υπολογισμοί για να καταλήξουμε σωστέ προτάσεις. Ε, ε εσείς που είχατε το θάρρος να μελετήσετε τις 780 τροπολογίες ε, βλέπετε ότι έχουμε ένα ζήτημα όσον αφορά την καταμερισμένη αρμοδιότητα. Επίσης το θέμα ότι ενδεχομένως αποφάσεις κατά πλειοψηφία ενισχυμένη πλειοψηφία θα πρέπει ε, να λαμβάνονται έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η δουλειά μας εδώ αλλά και στην ΕΜΠΕ, αυτό πρέπει να το ξέρουμε στην Ολομέλεια. Η κυρία Καστίγιο Βέρα από το ΕΛΚ και μετά... Ναι, Ωραία. Εξ ονόματο όμως ε, του ε, κυρίου Λάγκε, ο οποίο δεν μπορεί σήμερα να είναι εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσω το εξή, Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή αλλά και τους κοιόδης και φυσικά και τα άλλα μέλη της Επιτροπής μας ε, για τις προσπάθειές τους. Ε, μελέτησα τις ε, ε, πάνω από 700 τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και χαίρομαι διότι κάποιοι από τους προβληματισμούς που οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και η βιομηχανία είχαν υποβάλει προσεγγίζονται. Ε, υπάρχουν τροπολογίες τώρα οι οποίες αποτελούν ε, κατάλληλη ε, βάση για συζήτηση. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί πάντα προσπάθησε να εξεύρει προσέγγιση και συμβιβασμό, πράγμα όχι πάντα δύσκολο. Επίσης όσον αφορά τα benchmarks διαρκώς πρέπει να επικαιροποιούνται ε, και να λαμβάνονται υπόψη τα νέα στοιχεία. Οι εξελίξεις είναι καλές. Ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα είμαστε σε θέση να καθορίσουμε σωστές λύσεις ε, και να αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα των εκπομπών. Όσον αφορά τις λύσεις, πρέπει να πω ότι χαίρομαι γιατί αρκετές ε, πολιτικές ομάδες έχουν υποβάλει τροπολογίες οι οποίες στόχο έχουν την πιο δυναμική, πιο δυναμική κατανομή των ε, ορίων. Ε, Βεβαίω όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν χωρίς να δυσκολεύεται υπερβολικά η ζωή των μικρών επιχειρήσεων οι ίδιες ε, οι εταιρείες ε, μερικές φορές δεν ξέρουν καλύτερα μάλλον ε, είναι, ε, ποια είναι η καλύτερη λύση και μπορούν να πάρουν ε, αποφάσεις οι οποίες είναι, είναι πιο, πιο συμφέρουσες από πλευράς κόστους οφέλους. Ε, τέλος, όσον αφορά τις αντισταθμίσεις αποζημιώσεις, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιλέξουμε ένα πιο εναρμονισμένο και ίσο για όλους σύστημα. Ε, όσον αφορά την διαρροή ε, ε, άνθρακα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με μια καταποκοπήν αποζημίωση. Οι προτάσεις βέβαια οι οποίες έχουν υποβληθεί έχουν κάτι κοινό. Καμία από τις προτάσεις δεν βασίζεται σε ισχυρά ε, στοιχεία. Ε, οι περισσότερες ε, προτάσεις μπορεί να φαίνονται σωστές, αλλά όταν μιλάμε πλέον για συγκεκριμένα ποσοστά και όταν μπαίνουμε στις, στα πρακτικά στοιχεία εφαρμογής μιας τέτοιας προσέγγισης, εμείς σαν ΕΛΚ θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διαφορετικά στοιχεία έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την διαρροή του άνθρακα. Ε, επίσης, ε, ε, καλωσορίζουμε τη διαφοροποίηση μεταξύ δημοπρασιών και άλλων μορφών κατανομής. Ε, πρέπει πάντως να πω ότι ως ε, ΕΛΚ ε, εμείς θεωρούμε ότι φαίνεται, γνωρίζουμε ότι στο Συμβούλιο έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση όσον αφορά τις δωρεάν διανομές και ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ε, βρεθούν και κάποια αντικειμενικά ε, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και που θα εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας. Ο κύριος ε, ε, λέει, ο εισηγητής, από την αρχή είχε πει ότι ήθελε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και επομένως ε, θέλω να τονίσω ότι εάν θέλουμε να στεφθούμε από επιτυχία θα πρέπει οι συμβαστικές προτάσεις να ακολουθούν μια κοινή προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδης εισηγητής για την εξαιρετική εργασία που έχουν κάνει. Βεβαίω πρέπει να ανασκουμποθούμε και όχι μονάχα για να βρούμε συμβαστικέ λύσεις, αλλά και γιατί ε, ο χρόνος πιέζει. Έχουμε πέντε εβδομάδες έτσι ώστε να κλείσουμε τη θέση στην Ήτρε και μετά ε, οι συζητήσει θα είναι οπωσδήποτε πολύ έντονε. οπωσδήποτε θα χρειαστούμε μία ε, συνάντηση των σκιωδών ανά εβδομάδα και ίσω και δύο ανά εβδομάδα για τις τεχνικές ομάδε. Ένα μήνυμα λοιπόν θέλω να στείλω προς όλους. Πρώτα απ' όλα διαπιστώνουμε ότι η DG κλίμα δεν ξέρει και πολύ καλά. Ε, είναι λίγο όλα καλά και όλα ωραία και θαύμα όλα πάνε, αλλά δεν καταλαβαίνουν πολύ τις δυσκολίες, ενώ καταλαβαίνουμε ε, ότι τα προβλήματα είναι μεγάλα. Ε, το Think Tank Αγορά στις Βρυξέλλες 22 ε, Ιουνίου ε, ανέφερε ότι αυτό το Think Tank ότι είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές για το διοξίδιο του άνθρακα. Επίσης από την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει να βρεθούν πιο σοβαρές λύσεις τις οποίες όμως η DG Κλίμα τις βλέπει με πολύ μεγάλο δισταγμό όπως ας πούμε ε, οι διάδρομοι που αναφέρθηκαν προηγουμένως ο εισηγητής Ραντουγιέρ θεωρεί ότι ε, ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι για την γραμμική μείωση μέχρι το 2030 με την έννοια ότι δεν θα φτάσουμε ούτε καν ε, στα κάτω όρια των στόχων μας για την μείωση του διοξιδίου του άνθρακος. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο σύστημα ETS ε, και των εισαγωγών. 37,7 ε, ε, εκατομμύρια τόνοι μπήκαν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ. Εάν όμως δεν είχαμε τέτοιου είδους εισαγωγές χάλιβα, και ε, εάν ε, υπήρχε η δυνατότητα να επαναποληθούν ε, τα δικαιώματα βάσει του συστήματος ETS θα είχαμε μπορέσει να κερδίσουμε ένα δις. Από την άλλη πλευρά ισχυρή πίεση υπάρχει έτσι ώστε να έχουμε δωρεάν ποσοστώσεις. Αλλά εάν δώσουμε υπερβολικές ποσοστώσεις τότε θα μας πούν ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τη βιομηχανία. Στην αντίθετη περίπτωση θα ε, θα μας πούν ότι θα μας κατηγορήσουν ότι ε, ε, ε, ακριβώς απομακρυνόμαστε από τη βιομηχανία και δεν την θέλουμε. Ε, θα πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε κάποια στοιχεία πολύ σοβαρά υπόψη. Εάν εάν εξακολουθήσει να υφίσταται ε, ως έχει ε, αυτό το, το σύστημα της ε, διαρροής, τότε θα πρέπει να περάσουμε σε κάτι πιο δυναμικό. Θα πρέπει να ξαναυπολογιστούν τα benchmark βάσει της υφιστάμενης τεχνολογίας την φάση 4 κλπ. Επίσης θα πρέπει οπωσδήποτε να βεβαιωθούμε ότι αυτό το όφελος δεν θα πάει στις τσέπες των βιομηχάνων, αλλά γενικότερα στον τομέα και βεβαίως ε, θα πρέπει να είμαστε απολύτως διατεθειμένοι ε, και έτοιμοι να ε, να πληρώσουν τέλος πάντων ε, οι ε, παραβάτες ε, και νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε σωστοί θα πρέπει να ακολουθήσουμε είτε την θέση των πρασίνων σχετικά με τις αποζημιώσεις αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένει η decarbonization του ενεργειακού κλάδου για ορισμένο χρονικό διάστημα είτε να ακολουθήσουμε τη δική μας πρόταση. Επίσης ε, υπάρχει και η πρόταση για την ενεργειακή μετάβαση έτσι όπως έχει υποβληθεί ως πρόταση από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Τέλος, ε, μια και μιλάμε για το Ταμείο ε, της ε, Καινοτομίας, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όντως αυτό είναι ένα καλό εργαλείο στον δρόμο των δωρεάν ποσοστώσεων και αν βεβαίως θέλουμε να διατηρηθεί και η, ενεργεια, συγγνώμη, και η βιομηχανική βάση αλλά και να προστατευτεί το κλίμα. Επίσης, βλέποντας στο άρθρο 10 ε, γάμα, 10 C. Ε, η μόνη λύση που βλέπουμε είναι εμείς ως συν συνομοθέτες ε, να, είμαστε, να καθορίσουμε ε, σωστούς κανόνες που θα διασφαλίζουν ε, σωστές αρχές. Αλλά επί τη βάση αυτών των αρχών να αφήσουμε και τις χώρες να λειτουργήσουν μόνες τους τα συστήματα και όχι να αφήσουμε τα συστήματα αυτά στα χέρια των βιομηχάνων ή άλλων τέτοιων κατηγοριών ο κύριος Χένκελ, αντιπρόεδρος, ο οποίος ε, είναι και εισηγητής εξονόματος του ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φέντερ για το εξαιρετικό σας έργο. Από τη δική μου εμπειρία ως εισηγητή γνωρίζω ότι αγνοούμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας αφενός και τον παγκόσμιο χαρακτήρα του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Είναι πάντοτε δύο προβλήματα που έρχονται σε αντιπαράθεση. Τα θέματα της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων και της επαναβιομηχάνησης από την άλλη πλευρά. Δεν μιλάμε μόνο για διαρροή άνθρακα, αλλά και για διαρροή θέσεων εργασίας. Εγώ θα σας μιλήσω για δύο θέματα. Πρώτον, έχω την προσέγγιση της ε, ίσης κατανομής. Εγώ έχω εκφράσει την άποψη ότι ο στόχος για 50% δεν συμβαδίζει με τα στοιχεία στα οποία βασίζει η Κομισιόν την έκθεσή της. Οι Βέλγοι, λοιπόν, έχουν κάνει μια πρόταση η οποία αξίζει της προσοχής μας. 57% προς 43% η σχέση αυτή πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να δοθεί δυνατότητα για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το 57 προς 43 είναι μια αναλογία που είναι πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτή. Πιστοποιητικά που δεν χρησιμοποιούνται δεν θα πρέπει να πιστοποιούν, να δημοπρατούνται αλλά θα πρέπει να μεταφέρονται στην δωρεάν, την ελεύθερη κατηγορία. Νομίζω λοιπόν ότι αν, ακολουθήσουμε αυτή την οδό θα μπορούσαμε ακόμα και με μια αναλογία 55-45 να καταφέρουμε να συμβιβάσουμε αυτούς τους δύο στόχους της αντιμετώπισης του, της διαρροής άντρακα και της διαρροής θέσεων εργασίας. Και κάτι τελευταίο, ο εξυγχρονισμός ε, των διαδικασιών και της υποδομής θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών, όχι των ε, τραπεζών ούτε της Κομισιόν. Ο εκπρόσωπος των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να υπενθυμίσω τον βασικό στόχο αυτής της οδηγίας και του ETS. Η μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου σύμφωνα με την ε, απόφαση των Παρισίων. Θα πρέπει λοιπόν να απαλλαγούμε από τις ε, κρατικές επιδοτήσεις προς τα ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει λοιπόν για αυτό το σκοπό να, καταργηθεί το άρθρο 10 ο, με βάση το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τα ορυκτά καύσιμα. Ανεξάρτητες αναλύσεις έχουν αποδείξει ότι αντί να υπάρξει διαφοροποίηση, οι τρεις μεγαλύτερες ε, χώρες ε, στην ουσία ε, οι τρεις μεγαλύτεροι παραγωγοί ε, εκπομπών στην ουσία αξιοποιούν το σύστημα του ETS προκειμένου να αυξάνεται στο τέλος η χρήση του άνθρακα. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιούμε και να χρηματοδοτούμε παροχημένα συστήματα ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρηματοδοτεί συστήματα που θα είναι ε, συμβατά με τους στόχους τους περιβαλλοντικούς που έχουν τεθεί. Και αυτό θα πρέπει να, ε, σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσει ένα νέο ταμείο περιβαλλοντικής ανάπτυξης, μέσω του οποίου τα κράτη-μέλη θα λαμβάνουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του ενεργειακού του τομέα. Επίσης, δύσκολο θέμα θα είναι η αποζημίωση. Αυτή η αποζημίωση σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτελεί έναν μηχανισμό χρηματοδότησης των ρηπενόντων. Η γερμανική κυβέρνηση, για παράδειγμα, συμβάλλει, συνάπτει μάλλον συμβάσεις με εργολάβους μόνο εφόσον οι εργολάβοι αυτοί εκπέμπουν διοξίδιο του, του άνθρακα. 800 εκατομμύρια ευρώ έδωσε το 2013 έως το 2015 η γερμανική κυβέρνηση και θα συνεχίσει την ε, ίδια οδό έως το 2020. Χρειαζόμαστε να υπάρξουν λοιπόν κίνητρα μέσω της νομοθεσίας προκειμένου να ε, κινηθούμε σε μια ε, διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν στην οποία κινούνται αυτή τη στιγμή οι, τα κονδύλια και οι χρηματοδοτήσεις. Βεβαίως, αντί λοιπόν να δίνουμε ε, ενισχύσεις στους ρηπαίνοντες, η χρηματοδότηση θα πρέπει να κατευθύνεται σε τεχνολογίες απαλλαγής από τον άνθρακα προκειμένου να παραμείνει η Ευρώπη ανταγωνιστική στο περιβάλλον μετά την Συμφωνία των Παρισίων. Είναι σημαντικό η βιομηχανία λοιπόν να μπορέσει να χρησιμοποιήσει πλήρως αυτό το ταμείο, το νέο ταμείο καινοτομία το οποίο θα πρέπει να στηρίζει καινοτόμες ιδέες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρη την Ένωση. Εγώ προσβλέπω στη συνεργασία όλων των συναδέλφων και ελπίζω το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας να μην χάσουν αυτήν την ευκαιρία προκειμένου να συμβάλλουν με θετικό τρόπο στη θέσπιση αυτής της πολύ καινοτόμας νομοθεσίας. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, αρχικά ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον συνάδελφο του Φέντερ Λέι για τις συμβαστικές τροπολογίες που έχει καταθέσει. Όπως αντιληφθείτε και από τις τροπολογίες που καταθέσαμε εκ μέρους της ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, πρωταρχικός στόχος της αναθεώρησης του συστήματος είναι η μίση των εκπομπών για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το κλίμα και κατ' έκταση για ενίσχυση τη ποιότητα του των ανθρώπων. Και προ αυτή την κατεύθυνση είναι εμεί ζητάμε αυστηρότερα μέτρα για του μεγαλύτερου ρηπαντέ. Όσον αφορά τα δωρεάν δικαιώματα σε τομεί που κινδυνεύουν, τονίζουμε πω πρέπει να δίνονται με αναβαθμίσει και στοχευμένα με αυστηρά κριτήρια ώστε να υποφελούνται οι βιομηχανίε που έχουν πραγματικά ανάγκη. Πέραν του προβλήματο ε, ε τη διαρροή άνθρακα όμω, εξίσου σοβαρό ε, θεωρούμε εμεί ότι είναι και το πρόβλημα τη διαρροή θέσεων εργασία. Γι' αυτό τονίζομαι πως ιδιαίτερα τώρα εν μέσω οικονομικής κρίσης είναι σημαντικό να λάβουμε μέτρα για να στηρίξουμε τις μικρές βιομηχανίες, ιδιαίτερα στον Νότο, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία από και σημειώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά ενεργείας. Ε, διαφωνούμε λοιπόν με την ουσία της πρότασης που έχει κατατεθεί από την Κομισιό, καθώς οδηγεί στη δημιουργία ενός συστήματος εκπομπών που θα βοηθά τις μεγάλες βιομηχανίες που είναι κύριοι πέτοι των κλιματικών αλλαγών να αυξάνουν τα κέρδη τους σε βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας. Όσον αφορά το Ταμείο Εξυγχρονισμού, πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να έχουν σε αυτό συμμετοχή και λόγο εκπρόσωποι από όλα τα κράτη-μέλη και όχι μόνο από ορισμένα όπως προτείνεται. Μονάχα έτσι θα επιτύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων. Επίση, είναι σημαντικό το Ταμείο αυτό να στηρίξει τα κράτη-μέλη με κατακεφαλή ΑΕΠ 60% κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η πρόταση, αλλά με αναφορά όχι μόνο στο έτος 2013 όπως προτείνεται, αλλά και στα επόμενα έτη, το 2014 και το 2015. Λόγω της οικονομικής κρίσης και των δυσβάσταχτων μέτρων λιτότητας, πολλά κράτη-μέλη σημείωσαν μεγάλη μείωση τα τελευταία δύο χρόνια στο ΑΕΠ, και έχουν πραγματικά ανάγκη τη στήριξη από το Ταμείο Εξυγχρονισμού και νομίζω ότι είναι προφανές, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα τη της Ελλάδας. Ε, εμείς θα συμμετέχουμε σε συζητήσεις επικοδομητικά ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε όπου είναι δυνατό σε σημαντικές ε, ε, ε τροποποίησεις για να μπορεί να εκφραστεί κατά τον καλύτερο τρόπο η Επιτροπή της Ίντρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ. Mr. Dan Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Φέντερλε. Με 780 ανθρωπολογίες, καλή του τύχη. Να Σα ευχαριστήσω λοιπόν επειδή έχετε προσπαθήσει πραγματικά να συγκεντρώσετε τι καλύτερε ιδέε για την αναμόρφωση του συστήματος ε, εμπορία εκπομπών. Να πω τα εξή σχόλια. Σήμερα, κατά τη διάρκεια του μεσημερινού διαλύματο, είχαμε μια συνάντηση σχετικά με τον σχεδιασμό τη αγορά ηλεκτρική ενέργεια και σχετικά με την αύξηση των τιμών ενέργεια. Στην ε, αναθεώρηση και μεταρρύθμιση του συστήματο ETS, ε ακούσαμε κάποιου να κάνουν λόγο για αύξηση των τιμών ενέργεια. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει. Αν ισχύει αυτό, τι θα συμβεί με την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει ιδιαίτερος. Αλλά είναι περίπλοκα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται από την άλλη και με την ενεργειακή ένδυα. Μιλούμε τώρα για 50 εκατομμύρια Ευρωπαίους που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματο. Και αν αυξηθούν οι τιμές, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, θα φτάσουμε τα 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους όλα αυτά θα πρέπει κάπως να τα λύσει ο εισηγητή με τους κοιόδης μαζί και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πού ακριβώς θέλουμε να πάμε. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι αυτή η τιμή των 30 ευρώ ανατόνο διοξιδίου του άνθρακα που έχει ε, διακηρυχθεί ως ε, η χρυσή τομή θα έχει δύο επιπτώσεις. Πρώτον, η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντί να υποφεληθεί αυτή τη τιμή θα επιλέξει να μετακινηθεί, να μεταφερθεί στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω, κάπου θα πάνε. Και το δεύτερο και εξίσου προβληματικό είναι ότι μου φαίνεται μάλλον ύποπτο ότι έχουμε αυτή την τιμή των 30 ευρώ ανατόνο διοξιδίου του άνθρακα και ό του θαύματος αυτή είναι και η τιμή στην οποία καθίσταται εφικτό και σκόπιμο να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας. Τέλος πάντων, ελπίζω οι συνάδελφοι να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την ε, διάσωση και στήριξη της ε, βιομηχανίας και ε, προβληματίζει και το ζήτημα των καταναλωτών, πώς θα καταφέρουμε να τους προστατεύσουμε. Πολύ φοβάμαι ότι οι δυσκολίες θα εντείνονται δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ένα σχέδιο, αλλά κάποιο πρέπει να μα πει μέχρι πού θα φτάσουν οι τιμές ενέργειας και ποιος είναι ο στόχος τέλο πάντων. Θα στηρίξω όμω όσο μπορώ περισσότερο τον συνάδελφο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ήθελα να ε, συγχαρώ τον κύριο Φέντερ Λέι για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Θα αναφερθώ σε ένα ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκα και στις 13 Ιουνίου στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής και έχω υποβάλει και σχετική ερώτηση στις 27 Μαΐου. Και αυτό είναι η εξαίρεση της ελληνικής, ηλεκτροπαραγωγή της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής και κυρίως της ΔΕΗ, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, από τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε, ότι με βάση την οδηγία που συζητούμε, τη 2003 κάτω στο 87, τα κράτη-μέλη της Ένωσης, τα οποία έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερα από το 60% του μέσου όρου, με έτος αναφοράς του 2013, απαλλάσσονται από την υποχρέωση της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων. Ωστόσο η Ελλάδα, παρότι ξεπερνά ελαφρώς το κριτήριο αυτό το 2013, είχε 62%, εν λόγω του μνημονίου, πλέον για το 2014 έχει 59,7% του μέσου ε, κοινοτικού ΑΕΠ, άρα κάτω από το 60%. Και συνεχίζει η κατάσταση να είναι χειρότερη λόγω του μνημονίου και της οικονομικής κατάστασης. Αυτό λοιπόν που έχει σαν αποτέλεσμα σήμερα οι γειτονικέ χώρες της Ελλάδας, πλην της Ιταλίας, για πολλούς λόγους απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις να αγοράζουν ε, δικαιώματα. Πρώτα απ' όλα η Τουρκία δεν έχει τέτοια υποχρέωση, η Αλβανία δεν έχει τέτοια υποχρέωση, τα Σκόπια δεν έχουν τέτοια υποχρέωση και η Βουλγαρία έχει απαλλαγή. Τι έχει αυτό ως αποτέλεσμα. Η Ελλάδα να αναγκάζεται να κάνει αυξημένες εισαγωγές ρεύματος και αυτό να οδηγεί σε αυξημένα τιμολόγια. Και η ΔΕΗ να πληρώνει 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σας λέω κύριε Πρόεδρε επειδή το Σάββατο ήμουν στην Κοζάνη, σε μια περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί είναι πολλά εργοστάσια της ΔΕΗ που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα με λιγνίτη. Τα περισσότερα από αυτά, κύριε Πρόεδρε, βρίσκονται σε περιορισμένη λειτουργία. Και εισάγει η Ελλάδα ρεύμα από ένα εργοστάσιο που βρίσκεται στα Σκόπια, ενώ δίπλα, εντός των ελληνικών συνόρων και σε απόσταση 5 χιλιόμετρων, είναι ένα εργοστάσιο της ΔΕΗ το οποίο δεν λειτουργεί. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν πάει σφιχτεί αυτή η κατάσταση. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, θα σας δώσω και το υλικό να δείτε. Ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση από τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, από το Συνδικάτο Σπάρτακος, από την ε, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια αγωνία. Ποιο είναι το μέλλον της ΔΕΗ, τι θα γίνει, θα μπορέσει να ζήσει, θα μπορέσει να επιβιώσει. Μιλούμε για ενδεχόμενη απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Σας μεταφέρω λοιπόν κύριε Πρόεδρε και στους συναδέλφους και στον συνάδελφο την αγωνία των κατοίκων της περιοχής και ζητώ να γίνουν δεκτές δύο τροπολογίες που έχω καταθέσει. Η τροπολογία 548 και η τροπολογία 624. Και με αυτήν την τροπολογία, την 548, και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ζητούμε να ληφθεί υπόψη ως έτος βάσης και το 2014. Να μπορέσει να μπει και η Ελλάδα σε αυτή την εξαίρεση ήδη βρίσκεται σε μια άσχημη οικονομική κατάσταση με 1,5 εκατομμύριο ανέργους και να μπορέσει επίσης εάν ισχύσει αυτή η τροπολογία και η επόμενη, η 624, να πάρει τη δυνατότητα από το Ταμείο Εξυγχρονισμού για να στηριχθεί. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό και να έχουμε μια παρέμβαση στο ζήτημα αυτό και νομίζω ότι θα το δει θετικά και ο εισηγητή, θα το δει και η Επιτροπή. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, να σα μεταφέρω πραγματικά την αγωνία των χιλιάδων κατοίκων μια περιοχή στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαίδα, οι οποίοι αναμένουν από την Επιτροπή μα να του στηρίξει. Αυτή τη στιγμή, μόνο με τη λειτουργία του περιορισμού τη λειτουργία των εργοστασίων τη ΔΕΗ που έχουν το λιγνίτη, που είναι ε, μια δυνατότητα να παράγουν ρεύμα χωρίς εισαγωγές. Και αυτό είναι σημαντικό και για την ενεργειακή ασφάλεια. Δεν θα εξαρτώνται από εισαγωγές ρεύματος και είναι πολύ σημαντικό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την αγωνία εάν πραγματικά θα έχουν αύριο δουλειά. Μέχρι στιγμής έχουν χάσει 3.000 θέσει εργασία. Ελπίζω να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια και να μην κλείσει πραγματικά η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εμείς ευχαριστούμε, αγαπητοί συνάδελφε. Επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Τοσενόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλος αριθμός των τροπολογιών δείχνει πόσο πολύμορφο και περίπλοκο είναι το θέμα. Γι' αυτό άλλωστε έχουν γίνει τόσα χρόνια τόσες πολλές συζητήσεις. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι από εκείνους που πάντοτε τηρούσαν επιφυλακτική στάση απέναντι στο σύστημα. Πάντως είμαι σίγουρος ότι ο εισηγητής θα καταφέρει να καταλήξει στη συνεργασία με τους Σκιώδης σε μια λύση για να μην δημιουργηθούν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Και θέλω να αναφερθώ στο 10C και D. Στο 10C πρότεινα την αύξηση του ορίου στα 20 εκατομμύρια. Νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό προγραμμάτων. και θεωρώ ότι θα ήταν σωστό να καθοριστεί ένα κονδύλι 15 20 εκατομμυρίων. Για το 10D υπάρχει μια συμφωνία κυρίων μεταξύ των κρατών μελών που λέει ότι η επιλογή των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα των ε, ίδιων των κρατών μελών χωρίς την παρέμβαση από άλλα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτή η αρχή πρέπει να γίνει σεβαστή. Άλλωστε το Συμβούλιο έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι ο εισηγητής και οι σκιώδης θα μπορέσουν να καταλήξουν σε μια αξιοπρεπή λύση ε, προκειμένου και εμείς από την πλευρά της Επιτροπής μας να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην όλη συζήτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπλάνκο Λόπες. Πολλά είναι τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν εδώ, αλλά εγώ θα ήθελα ε, να ασχοληθώ με το θέμα της αποζημίωσης των εμέσων ε, κοστών ε, συνδεδεμένων με την ε, με την διαρροή άνθρακα. Ε, μέσω της τροπολογίας μου 488 ε, προτείνω ένα σύστημα εναρμονισμένης αποζημίωσης. Εγώ ορίζω το ποσοστό στο 3%, η ομάδα μου 2%, στην τροπολογία 217, άλλοι δε αυξάνουν το ποσοστό μέχρι το 19%, ε, βάσει της τροπολογίας 222 μαζί με κάποιους άλλους μηχανισμούς αποζημίωσης. Είναι βέβαιο ότι το έτος 2015 περισσότερα από 450 εκατομμύρια ευρώ ε, δόθηκαν, σπαταλήθηκαν ε, στην κάλυψη των, της αντιστάθμισης των εμέσων κοστών, πράγμα που όμως οδηγεί εν τέλει σε αθέμητο ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία βιομηχανία. Πρόκειται για ένα θέμα ε, επί της οποίας ε, καλώ τον εισηγητή να βρει ευρεία συνένεση και συμβιβασμό. Ε, αυτό είναι σημαντικό και για την σχέση μας με την Επιτροπή Περιβάντος αλλά και για τις περαιτέρω σχέσεις μας με την Κομισιόν και το Συμβούλιο και τις μελλοντικέ μας συζητήσεις με αυτά τα όργανα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν έχει ζητήσει κανεί άλλο τον λόγο. Να προσθέσω μερικά σχόλια, αν με επιτρέπετε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Σα ευχαριστώ, Φρέντερικ, για την πολύ δουλειά που έχει κάνει. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο σε τέτοιε περιπτώσει ε, να πληρώσει όλε τι προσδοκίε μα. Αυτό είναι βέβαιο. Όμω, βλέπουμε ότι κάποιε από τι τροπολογίε που έχουν κατατεθεί δεν ελήφθησαν υπόψη. Πολύ σοβαρά τουλάχιστον. Και θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που ανέφερε και ο συνάδελφος Τωσενόφσκι και κάποιοι άλλοι. Οι τροπολογίες που αφορούν το άρθρο 10C και 10D. Γιατί εμείς βεβαίω θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας ε, για το κλίμα μέχρι το 2030, όμως έχοντας κατά νου και την ευρωπαϊκή βιομηχανική μας και οικονομική μας ανταγωνιστικότητα. Είναι σκοπός αυτός της, ε, και αρμοδιότητα τη ΣΥΤΡΕ. Θέλουμε λοιπόν τον πιο αποτελεσματικό δυνατό μηχανισμό αποζημίωση και προκειμένου και οι οικονομίες ε, με υψηλής κατανάλωσης ε, άνθρακα να εξυγχρονιστούν. Δεύτερον, θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα ίσο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ χωρών με διαφορετική αφετηρία στην ενεργειακή αυτή μετάβαση. Γιατί κάποιε χώρε ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια, ενώ κάποιε πριν από 8, 10, 12 χρόνια. Δεν είναι το ίδιο. Και τρίτο θέμα, θέλουμε να μετριάσουμε τυχόν αρνητικό αντίκτυπο του εξυγχρονισμού προ του καταναλωτέ. Και θέλουμε και μια γενική αναθεώρηση, μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού ETS, ε, απλουστευμένη διακυβέρνηση, τεχνολογική ουδετερότητα, ευελιξία στην αλλαγή και στην τροποποίηση των ρυθμιστικών κανόνων. Βεβαίως, ε, προβλεψιμότητα μακροπρόθεσμα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Επομένω, τονίζω και πάλι τα άρθρα 10C και 10D είναι πολύ σημαντικά για μας. Το ανέφεραν και κάποιοι συνάδελφοι, γιατί από κοινού καταθέσαμε ορισμένε τροπολογίε. Είναι πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε εδώ το περιεχόμενο των ε, διατάξεων, αν έχουμε κατά νου ε, την οικονομική ανταγωνιστικότητά μας. Παρότι κατανοώ ότι δεν είναι εύκολο αυτό για τον εισηγητή. Η κυρία Γκοστέτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήμουν σε μια άλλη επιτροπή, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Όμως χαίρομαι πολύ που κατάφερα να έρθω έστω και καθυστερημένα. Με τα χαράς άκουσα τα όσα είπατε και συμφωνώ απολύτως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Επιτροπή μας, την Ήτρε, πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα της ε, βιομηχανίας μας. Λέει ο πρόεδρος, υπάρχουν προβλήματα με τη δερμηνία, όχι εξ όσων γνωρίζουμε, σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. αν θέλετε να ξεκινήσετε από την αρχή, λέει ο Πρόεδρος. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν θα ξεκινήσω την αρχή. Απλώ θέλω να πω ότι συμφωνώ μαζί σα, γιατί στην Επιτροπή Βιομηχανία είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι στην Ευρώπη θα έχουμε μια βιομηχανία που θα διατηρήσει ε, την διεθνή τη ανταγωνιστικότητα για να εξακολουθήσει να δημιουργεί θέσει απασχόληση και ταυτόχρονα είναι και μοχλό ε, καινοτομία ε, για την απομάκρυνση από τον άνθρακα. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν αυτή την ισορροπία μεταξύ των δύο στόχων. Πώ θα τα καταφέρουμε τώρα μαζί με αυτή την αγορά του άνθρακα, ούτω ώστε το κόστο του άνθρακα να μην ε, τιμωρεί εντό αγωγικών ε, τις επιχειρήσει, ε, θα καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τη τιμή του άνθρακα για να κάνουμε το πέρασμα ε, σε μια νέα, νέα οικονομία μακριά από τον άνθρακα, πώς θα δώσουμε κίνητρα στις δικές μας επιχειρήσεις σε σχέση με άλλες, παρότι ήδη ε, συμμορφούνται με πρότυπα πιο αυστηρά σε σχέση με άλλες περιοχές. Είναι περίπλοκο λοιπόν το ζήτημα πρέπει να δοθούν ισχυρές και ισορροπημένες ε, απαντήσεις, δίνοντας ένα περιθώριο ευελιξίας ό,τι αφορά ε, τον συντελεστή διόρθωση, τον μη κλαδικό θα μπορούσαμε να τον προβλέψουμε και να έχουμε και ένα benchmarking ανάλογα με τις πραγματικές τεχνολογικές εξελίξεις και σε όσους ε, είναι πραγματικά εκτεθειμένοι να δίνουμε αντίστοιχες ποσοστώσεις. Πρέπει να έχουμε και πιο δυναμικές ποσοστώσεις και δικαιώματα εκπομπών και να αποφύγουμε το πλεόνασμα των ε, αδικαιολόγητων ε, δικαιωμάτων εκπομπών. Και για το μη ETS επίσης ε, κλάδο θα πρέπει να γίνει λόγος γιατί θα συμμετάσχει στο όλο σύστημα και γι' αυτό περιμένω με ανυπομονησία τις προτάσεις της Κομισιόν που λογικά θα λάβουμε την επόμενη εβδομάδα. Αυτά είχα να πω. Φαντάζομαι συνεχίζω στο ίδιο πνεύμα με τις δικές σας παρατηρήσεις προηγουμένως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τη Γενική Διεύθυνση Κλίμα. Μέρη Βερόνικα Τόσακ Πετέρσκι. Εκπροσωπεί η Γενική Διεύθυνση Κλίμα. Διευθύντρια, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και σας ευχαριστώ και όλους για την τόσο ενδιαφέρουσα και πλούσια αυτή συζήτηση. Δεδομένα του αριθμού των τροπολογιών, είναι σαφής η σημασία αλλά και το ενδιαφέρον ε, που συγκεντρώνει το ETS και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό. Θα ήθελα να ε, σταθώ στις τρεις κύριες πτυχές του ζητήματος. Καινοτομία, αλληλεγγύη και δύο λόγια και για το διοικητικό άκθος. Πρώτον, να πω και πάλι ότι μελετήσαμε τις τροπολογίες, παρακολουθήσαμε και σήμερα τη συζήτηση και βλέπουμε ότι πολλές τροπολογίες αφορούν με κάποιον τρόπο την καινοτομία. Με ενδιαφέρον σημειώνω εδώ τον προβληματισμό για την αύξηση της, ε, ε της χρηματοδότησης για συγκεκριμένα καινοτόμα προγράμματα και ότι πρέπει να δοθεί καθοδήγηση για το πώς θα πρέπει να εξολογούνται αυτά τα προγράμματα για να γίνονται περαιτέρω συζητήσεις για την κατάλληλη ισορροπία επιμερισμού του κινδύνου ε, όπως αυτό εκφράζεται και με την χρηματοδότηση. Ήθελα να επισημάνω ορισμένα απλώ ε, σημαντικά ζητήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τρόπο με τον οποίο επικαιροποιούνται τα benchmarks είναι εξίσου σημαντικό για την ε, σκοπιά τη ε, καινοτομία. Το έχω πει ήδη σε αυτή την επιτροπή, δεν θέλω να τα επαναλάβω, όμω το πλαίσιο της, καταποκοπήν ε, ποσού για τα benchmarks ε, δίνει μια καλή ισορροπία και για τα επίπεδα φιλοδοξίας μας, αλλά και για να προστατεύσουμε τους ε, κλάδους που κινούνται με μεγαλύτερη καθυστέρηση. Και έχουμε δει πολλά σχόλια και από αυτή την άποψη. Δεύτερον, για τους μηχανισμούς αλληλεγγύης. Ταμείο Εξυγχρονισμού, άρθρο 10C και 10% ανακατανομής. Ήθελα να επαναλάβω ότι αυτά τα στοιχεία αλληλεγγύης ήταν θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη συνένεσης μεταξύ των αρχηγών και των κυβερνήσεων για να υιοθετηθεί ο στόχος του τουλάχιστον 40% τον Οκτώβριο του 2015. Ε, και τα όσα υπόθηκαν σήμερα το απόγευμα για την ε, την πρόκληση των επενδύσεων ε, που ε, συνεπάγεται αυτό που λέμε για τις ε, χώρες με χαμηλότερο εισόδημα. Έτσι, οι μηχανισμοί αλληλεγγύης είναι πολύ σημαντικοί και για την επίτευξη των στόχων. Δεν θέλω να περάσω σε όλες τις λεπτομέρειες της πρότασης που έχει τεθεί επιτάπητος για το 10Γ, τονίσω μόνο ότι θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση των μηχανισμών που θα αυξήσουν τη διαφάνεια, ιδίω ό,τι αφορά τι δημοπρασίε, ε, και αυτό θα έχει και μεγαλύτερη περιβαλλοντική αξία. Τώρα, το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Πολύ σημαντικό είναι να έχουμε κατά νου τον ε, κυρίαρχο στόχο να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα που θα ε, πραγματοποιούνται με βάση αυτό τον μηχανισμό θα διευκολύνουν τον πραγματικό αυτό εξυγχρονισμό της βιομηχανίας και πάντα σε διαφανή βάση. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που συνδέονται με το μέγεθος, τη σύνθεση, Και εδώ πρέπει να έχουμε κατά νου τον βασικό αυτό στόχο. Τελευταία μου παρατήρηση για το διοικητικό άκθος. Νομίζω πολλές φορές έχω ακούσει αυτή την ε, Επιτροπή στη συζητήση για το νέο ETS ε ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για την ε, μείωση του διοικητικού άχθους. Θα ήθελα και εγώ να έχουμε κατά νου αυτόν τον στόχο όταν εξετάζουμε τροπολογίες για αυτή την νομοθετική πρόταση. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω ότι κάποιες τροπολογίες αντιβαίνουν απολύτως ε, στην αρχή αυτή του περιορισμού του διοικητικού άχθους. Για παράδειγμα, ο επανυπολογισμός των benchmarks από την αρχή, πριν την αρχή της ε, τέταρτης περίοδου. Ή ε, κάθε δύο χρόνια να γίνεται η ε, ελεύθερη κατανομή. Η κατανομή ελεύθερων δικαιωμάτων. Μπορούμε να βρούμε και, άλλες, άλλα παραδείγματα, διεύρυνση πεδίου εφαρμογή για τις ε, εδώ είμαστε για να σας ακούσουμε. Όμω θα πρέπει όλα αυτά να βαίνουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, να είναι στοχευμένα, με σκοπό τον εξυγχρονισμό ε, του ενεργειακού κλάδου. Θα ήθελα όμως να πω ότι οι τελικές επιλογές θα πρέπει ε, να τηρούν και τις αρχές ε, της καλύτερης νομοθεσίας. Δεν ήθελα να μακρηγορήσω. Βεβαίως, αν θέλετε περαιτέρω διευκρινήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Να επαναλάβω μόνο ότι είμαστε διατεθειμένοι όλα αυτά να τα συζητήσουμε περαιτέρω και βεβαίως θέλουμε να καταλήξουμε σε μία ε, άρτια πρόταση για αυτόν τον πολύ σημαντικό φάκελο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιγητά. Φρέντερικ Φέντερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η συζήτηση που μόλις προηγήθηκε καταδεικνύει και τη σημασία του θέματος αλλά και τις ε, διάφορες ε, απόψεις που εκφράζονται. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας και τη βιομηχανική αλλά και όλες τις άλλες διαστάσεις του θέματος. Γνωρίζουμε ότι πολλοί κλάδοι της οικονομίας ε, ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Κάποιοι θέλουν να κινηθούμε σε μία κατεύθυνση, κάποιοι άλλοι να κινηθούμε σε κάποια διαφορετική διάσταση, κατεύθυνση. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την περιφερειακή διάσταση και η συνάδελφος ε, μας έδωσε και συγκεκριμένα ε, παραδείγματα για το πώς το ETS επηρεάζει την καθημερινή ζωή των πολιτών στη φορολογία και αλλού. Επίσης θα λάβουμε υπόψη μα το έργο της Κομισιόν, την οποία και ευχαριστώ παρά γιατί για όλη τη συνεργασία της, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές ε, έχουμε διαφορετικές απόψεις και με το Συμβούλιο ισχύει το ίδιο. Έχουμε λοιπόν πολύ δρόμο μπροστά μας. Ένα θέμα που αναφέρθηκε, η κυρία Γκροστέτ νομίζω το είπε. Είναι εκείνη που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ποιοι είναι τελικοί, τελικώς αυτοί που διατρέχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, θα γίνουν έντονες συζητήσεις και στο τέλος θα καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς. Και αυτό είναι αναγκαίο γιατί αν δεν καταφέρουμε εμείς να καταλήξουμε εδώ σε αυτή την Επιτροπή δεν θα μπορέσουμε να πάμε ούτε στην Επιτροπή Ένβη. Ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για τη συζήτηση. Αύριο θα έχουμε την πρώτη συνεδρίαση σκιονδών. Ε, θα γίνουν πάρα πολλές συνεδριάσεις βέβαια το επόμενο διάστημα, όπως είπε και ο συνάδελφος. Σε κάθε περίπτωση εγώ δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Αγαπητοί φίλοι, αύριο στις 5 το απόγευμα κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ήτρε και Κούλτ για τις, τους δημιουργικούς κλάδους πολύ σημαντική συνεδρίαση. Εγώ σε μια ώρα φεύγω για Μπρατισλάβα ως πρωτεύουσα της χώρας που έχει την Προεδρία. Αλλά θα έχω επιστρέψει μέχρι αύριο, ελπίζω πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, της κοινής συνεδρίασης αυτής που θα κάνουμε με την Επιτροπή Πολιτισμού. Ο κύριος Ρούμπικ, επειδή είναι το παλαιότερο μέλος, είναι νέος βέβαια, αλλά είναι το παλαιότερο μέρος, μέλος της Επιτροπής μας. Είναι μέλος εδώ και 17 χρόνια της Επιτροπής Ήτρε. Εκείνος λοιπόν θα προεδρεύσει τη συνεδρίαση αύριο στις 5 το απόγευμα. Και εγώ θα τρέξω να βιαστώ για να γυρίσω όσο το δυνατόν νωρίτερα. Κύριε Φέντερλη, επειδή είναι η τελευταία μας συνεδρίαση για φέτος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βοηθούς, τους συμβούλους των πολιτικών ε, ομάδων, τους υπαλλήλους της Επιτροπής Ήτρε, τους συναδέλφους για την συνεργασία που είχαμε και θα ήθελα κύριε Μπούζεκ να ευχαριστώ εσάς, να ευχαριστήσω προσωπικά εσάς για το έργο σας. Είπαμε και στους συντονιστές σήμερα ότι εμείς έχουμε πολύ συχνά τα δικά μας θέματα, ερχόμαστε, φεύγουμε, αλλά ο πρόεδρος είναι πάντοτε εδώ σας ευχαριστώ για όλη σας τη στάση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Αυτά είχα σκοπό να πω εγώ όμως αύριο στις 6.30. Αν καταφέρω να γυρίσω από την Πρατισλάβα. Παρόλα αυτά, αύριο συνεδρίαση με προεδρεύοντα τον κύριο Πολ Ρούμπικ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.